Σας χαιρετίζω λοιπόν εδώ και πάλι και αρχίζω και πάλι τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ελπίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι αναπαυμένοι ε, έχουν επανέλθει. Έχουμε εδώ επισκέπτες συγκεκριμένα τον Υπουργό για Γεωργία, Φυσικούς Πόρους και Περιβάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Προεδρίας. Είναι ο κύριος Σοφοκλής Αλετράρης. Το Σαββατοκύριακο το είχα πάει στην Κύπρο. Συνεδρίασε το άτυπο συμβούλιο και γύρισα πλήρης ενθουσιασμού γιατί άκουσα συγκεκριμένα στοιχεία στο περιεχόμενο της Προεδρίας και ξέρω ότι ο κύριος Σοφοκλής Αλετράρης είναι η Δήμων σε θέματα πολιτικής υδάτων. Είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της Προεδρίας. γιατί το θέμα των υδάτων, η ποιότητα του υδάτος δεν αφορά μόνο τον νότο της Ευρώπης. Είναι κάτι που αφορά όλη την Ευρώπη και πρέπει να μας απασχολήσει στην ομοθεσία μας. Υπάρχει η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και ένα άλλο συγκεκριμένο θέμα που συζητήθηκε ήταν πώς θέλουμε να υπάρξουν μέτρα προσαρμογής για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα μέτρα αυτά. Γιατί όπως είναι γνωστό, όταν αρχίζουμε να μιλάμε για λεφτά, σταματάνε οι φιλίες. Αυτό ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τον Υπουργό εδώ. Καλώς ήρθατε αγαπητέ φίλε και καλωσορίζω το εξάμεινο της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, όχι μόνο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τον ένα από τους πυλώνες του οικοδομήματος κρατών, θεσμών, οργανισμών ιδεών, νομοθετημάτων και πολιτικών που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανάφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εναρκτήρια ομιλία του, η κοινοτική μέθοδος να επιλύονται δηλαδή οι διαφωνίες με το διάλογο και τη συνένεση αποτελεί τη ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκομαι έτσι εδώ και γιατί προέρχομαι από μια χώρα στην οποία οι δημοκρατικοί θεσμοί και ο διαχωρισμός των εξουσιών λειτουργούν υποδειγματικά στην οποία το πολιτικό σύστημα αλλά και η σύνθεση του εκλογικού σώματος είναι τέτοια ώστε μόνο μέσα από διάλογο, συμβιβασμούς, φυσικά όχι σε θέματα αρχών, και αλληλοκατανόηση μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας μπορεί να διαμορφώσουν πολιτικές νομοθετήματα που να αντιπροσωπεύουν τις εύλογες προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δώσατε να βρεθώ σήμερα μαζί σας και να σας ενημερώσω αλλά και για να σας ακούσω για ένα πάρα πολύ σημαντικό πυλώνα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό του περιβάλλοντος. Το κοινοτικό κεκτημένο για θέματα περιβάλλοντος καθορίζει την πορεία της Ευρώπης προς την αηφορία. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ακολουθία και συμβατότητα των δημοσιονομικών και οικονομικών ενεργειών με τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφόρο ανάπτυξη. Η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι δεν θα αποβούν μακροπρόθεσμα σε βάρος του περιβάλλοντος οι σημερινές προτεραιότητες για τη λήψη βραχυπρόθεσμων δράσεων σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι η σημερινή κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί και ως ευκαιρία για νέες πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί η αποστολή βασικού μηνύματος πολιτικής από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Εαρινό Συμβούλιο του 2013 με στόχο το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με βάση και την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου θα γίνει συζήτηση πολιτικής για το θέμα αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο, μια από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι να εργαστούμε προς μια περισσότερο αποδοτική και εφόρο Ευρώπη. Μέσα από τις δραματικές συνέπειες του τωρινού έντονα μεταβαλλόμενου και ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, αναδείχθηκε και η ανάγκη για στοχευμένες προσεγγίσεις για την επίτευξη αεφόρου ανάπτυξης. Πιστεύω ότι το κοινό μας όραμα της διάσκεψης του Ρίο, έστω και αν δεν ικανοποιεί πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την αηφόρο ανάπτυξη στο επίκεντρο των εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προτεραιοτήτων. Τώρα η κοινή πρόκληση για όλους είναι να προωθήσουμε όλα όσα συμφωνήθηκαν και να διασφαλίσουμε ουσιαστική δράση για φόρο ανάπτυξη, πράσινη οικονομία και εξάλληψη της φτώχειας. Τα αποτελέσματα του Ρίο θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος με στόχο την έγκριση συμπερασμάτων για την περαιτέρω εξειδίκευση των επιδιώξεων και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε διεθνές επίπεδο, στη Νέα Υόρκη, στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που υιοθετήθηκαν και η ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαβουλεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης των στόχων αηφόρου ανάπτυξης καθώς και του διεθνούς θεσμικού πλαισίου. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να συνεχίσει να πρωτοστατεί και να παραδειγματίζει τις κοινέ προσπάθειες της ανθρωπότητας για την αντιμετώπιση των αλληλένδετων περιβαλλοντικών κρίσεων της εποχής μας η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή βήματα και συνέδρια. Στον ευρύ τομέα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της διαφύλαξης των νερών και της κλιματικής αλλαγής. Παρόλο που το νερό είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την εφόρο ανάπτυξη, τα νερά της Ευρώπης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλές απειλές. Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ανατρέψει την φυσική ισορροπία που υπήρχε. Παρά τη σχετική νομοθεσία και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αεφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων των προεδριών. Όπως γνωρίζετε, στο στάδιο αυτό βρίσκεται υπό διαμόρφωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το οποίο θα επιδιωχθεί μεταξύ άλλων να ολοκληρωθούν οι σχετικές πολιτικές. Για το σχέδιο αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος πρόταση για συμπεράσματα Συμβουλίου. Ήδη προηγήθηκε διάλογος στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκοσίας που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σαββατοκυριακό και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη δική του συνεισφορά. Ενώ θα συγκληθεί τον Νοέμβριο συνέδριο για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το σχέδιο. Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί επίσης για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας στα νερά. Επιδίωξή μας είναι να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωκοινοβούλιο. Για το θέμα άρχισαν ανεπίσημες επαφές. Εάν βέβαια αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα επιδιώξουμε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο του Δεκέμβρη. Έρχομαι τώρα στο μεγάλο θέμα της κλιματικής αλλαγής οι επιπτώσεις από την οποία αναμένεται να είναι σε τέτοια έκταση την οποία δεν αντιμετώπισε η ανθρωπότητα στη σύγχρονη ιστορία. Παραλάβαμε από τη Δανία τη σκητάλη του δρόμου προς την Τόχα και θα δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό για την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης. Τον Οκτώβρη το Συμβούλιο θα υιοθετήσει συμπεράσματα σχετικά με τις διαπραγματευτικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου που πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί. Η συνετή εφαρμογή και βελτίωσή του μπορεί να ενισχύσει και τις ευρωπαϊκές προπτικές για οικονομική ανάπτυξη. Ο δρόμος προς τα εμπρός θα εξεταστεί μετά την σχετική έκθεση της Επιτροπής. Σε περίπτωση που αυτή υποβληθεί πριν από το τέλος της Προεδρίας της Κύπρου, θα προωθήσουμε το θέμα κατάλληλα. Θα εργαστούμε επίσης για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σε δύο θέματα που βελτιώνουν την κοινοτική πολιτική και μπορούν να συνδράμουν θετικά στον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αναφέρομαι στην αναθεώρηση του συστήματος παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε μεταξύ άλλων να αντικατοπτρίζει τις μέχρι τώρα εμπειρίες καθώς και τη συμπερίληψη του τομέα των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήση γης και τη δασοκομεία στις δεσμεύσεις για μείωση των ολικών εκπομπών. Η ενσωμάτωση της προσαρμογής στην αλλαγή κλίματος στις άλλες πολιτικές θα έχει την υποστήριξη της Προεδρίας της Κύπρου. Μαζί με το νερό και το θέμα αυτό απασχόλησε το άτυπο Συμβούλιο του Ιουλίου με έμφαση στη χρηματοδότηση που θα πρέπει να στηρίξει την στρατηγική που τώρα ετοιμάζεται. Επίσης, σε περίπτωση που θα κατατεθούν έγκαιρα οι προτάσεις για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από ελαφρά οχήματα και ελαφρά επαγγελματικά καθώς και για τα φθουρούχα αέρια θα προωθηθεί η παρουσίασή τους από την Επιτροπή και πιθανό μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις είναι αυτό της προστασίας και διαχείρισης της βιολογικής ποικιλότητας παρά την πλούσια ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές πολιτικές, συνεχίζουμε να, συμπεριφερόμαστε έως αν το περιβάλλον να κατέχει μια απεριόριστη ικανότητα να παράγει, να προσαρμόζεται στις μία εφόρες καταναλωτικές μας συνήθειες και να δέχεται και απορροφά τα απόβλητά μας. Στον εξαιρετικά σημαντικό αυτό τομέα θα γίνουν διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για την Βιολογική Ποικιλότητα τον Οκτώβριο του 2012 στην Ινδία. Η Προεδρία θα διασφαλίσει την ουσιαστική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις και τις μετέπειτα ενέργειες, στηριγμένη στα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στο στρατηγικό σχέδιο την κινητοποίηση πόρων, την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και στη θαλάσσια ιοπικιλότητα. Η Προεδρία της Κύπρου θα ετοιμάσει επίσης συμπεράσματα για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Παράλληλα, θα ενεργήσουμε κατάλληλα όσον αφορά την αναμενόμενη νομοθετική δέσμη για την εφαρμογή του πρωτοκόλου της Νακόια για την πρόσβαση και τη συμμετοχή στα ωφέλη από τους βιολογικούς πόρους, ανάλογα πάντα με το χρονικό στάδιο της υποβολής της. Προχωρώντας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, δυστυχώς αυτός εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση αφού η ένταση στη χρήση των πόρων και η δημιουργία αποβλήτων δεν έχουν αποσυνδεθεί από το ρυθμό της κοινωνικής ανάπτυξης. Η Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία στην πρόταση για τη διάλυση των πλοίων σε ασφαλείς και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις. Στο Συμβούλιο του Οκτώβρη θα διεξαχθεί συζήτηση ανατολισμού σχετικά με την πρόταση να τεθεί τέρμα στην εξαίρεση από την απαγόρευση του καδμίου στις μπαταρίες σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία, αρχική μας επιδίωξη ήταν η επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Σε περίπτωση φυσικά που θα διαφοροποιεί του το χρονοδιάγραμμα εξέτασης του θέματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ των πραγμάτων, θα προχωρήσουμε τώρα σε προσπάθεια επίτευξης Γενικής Συμφωνίας στο Συμβούλιο Οκτωβρίου. Η Προεδρία θα είναι επίσης έτοιμη να χειριστεί μερικά άλλα σημαντικά θέματα οριζόντιας εμβέλειας. Μεταξύ αυτών, εξέχουσα θέση έχει η πρόταση για το νέο κανονισμό LIFE με προτινόμενο προϋπολογισμό 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε μέχρι τώρα, δεν έγινε δυνατή η επίτευξη μερικής πολιτικής συμφωνίας. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε τις συζητήσεις όσο το δυνατό περισσότερο και να εισέλθουμε σε τριλόγους παράλληλα με την πρόοδο στις άλλες τομεακές προτάσεις ώστε να έχουμε συμφωνία πάνω στον κανονισμό μέχρι το 2013. Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να καθορίσει μια νέα περιβαλλοντική στρατηγική προς την πράσινη οικονομία υπό το φως των συμπερασμάτων του Ιουνίου του 2012 των αποτελεσμάτων του Ρίο και της ανακοίνωσης για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Προκαταρκτικά, προγραμματίστηκε παρουσίαση του προγράμματος από την Επιτροπή στο Συμβούλιο Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που υπάρξει αντικείμενο, τότε θα ετοιμαστεί έκθεση πρόοδου. Ένα άλλο θέμα προτεραιότητας για την Προεδρία είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με στόχο να βελτιωθούν οι διαδικασίες και η ποιότητα των μελετών. Ανάλογα με το στάδιο της δημοσίευσης της πρότασης, η Προεδρία θα προωθήσει το θέμα όσο το δυνατό περισσότερο. Στοχεύομαι σε συζήτηση ανατολισμού ή έκθεση πρόοδου στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έντιμοι ευρωβουλευτές δεν έχουμε ψευδεσίσεις για το ότι η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά από μια μικρή σε έκταση και πληθυσμό χώρα θα δοκιμάσει τις δυνατότητές μας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, ιδιαίτερα στα θέματα περιβάλλοντος, όπου οι θεσμοί, οι νομοθεσίες και οι μηχανισμοί βρίσκονται σε συνεχή μετασχηματισμό. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις αυτές, έγιναν διευθετήσεις ώστε να διασφαλιστεί στο μέτρο του εφικτού η ορθολογική διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας. Δεν θα σας απασχολήσω με λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να σημειώσω μερικά σημαντικά κατά την άποψή μου σημεία. Πρώτον, για τα θέματα της εφόρου ανάπτυξης και άλλα διεθνή θέματα γενικής φύσεως, έμπειρα στελέχη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας ήδη στηρίζουν τους Κύπρους εκπροσώπους στις διάφορες συναντήσεις. Δεύτερον, άλλα διεθνή θέματα όπως η βιολογική ποικιλομορφία και η διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπανση καλύπτονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δανίας με συμφωνία ανάθεσης. Διατηρούμε φυσικά την πολιτική ευθύνη και σε συναντήσεις υπουργικού επίπεδου ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, λόγω της μεγάλης του σημασίας και παρά την πίεση που θα ασκηθεί και στην ηγεσία του Υπουργείου και το προσωπικό, αποφασίστηκε ότι το πολύπλοκο θέμα των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα το χειριστεί κυπριακή ομάδα ενισχυμένη με μερικούς ξένους εμπειρογνώμονες. Κύριε Πρόεδρε, οι μέχρι τώρα συναντήσεις μου με και αρκετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου επέτρεψαν να διαπιστώσω την ύπαρξη κοινού πιστεύω για συνεργασία, πνεύματος κοινού μέλλοντος, αλληλοεκτίμησης και επιθυμίας να ακούσει ο ένας τον άλλο. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλές ευκαιρίες να διαπιστώσουμε το πνεύμα αμοιβιότητας και αλληλοσεβασμού που χαρακτηρίζει όλα τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είμαι αισιόδοξο για την έκφαση της Προεδρίας μας. Θα εργαστώ ώστε μαζί να συνεχίσουμε να χτίσουμε και να διαμορφώνουμε το μέλλον της Ευρώπης απερίσπαστη από την έντονη πίεση για τη διαχείριση κρίσεων ενεργώντας για δράση με συλλογική σοφία. Αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου θα καθοδηγούμε από τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. Αλλά δεν θα είμαι ένας ουδέτερος θεατής. Τις εβδομάδες και τους μήνες που έρχονται θα αναζητήσω κοινό έδαφος με όλους με τη λογική με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και η μετριοφροσύνη και η ταπεινότητα που μου προκαλεί το δέος για το όλο εγχείρημα. Γνωρίζω ότι I have promises to keep and miles to go before I sleep. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε και την υπομονή που είχατε να με ακούσετε. Τώρα είναι η σειρά μου να σας ακούσω και να σας απαντήσω στο βαθμό φυσικά που γνωρίζω και που μπορώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας αυτή, για την παρουσίαση του προγράμματός σας. Είναι αυτά που αναμέναμε για το προσεχές ε, εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας και η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της ε, Προεδρίας όπως την παρουσιάσατε. Είναι πολύ καλό να μην ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας, αλλά να βλέπουμε και ε, προς το Ρίο είναι η μεγάλη συνδιάσκεψη. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη έχει μια διεθνή ευθύνη για το πώς θα δράσουμε για μια καλύτερη παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, για μια, ένα πιο δίκαιο κόσμο και για την προστασία του κλίματος. Οπωσδήποτε το αναφέρετε κι εσείς. Παραδοσιακά τώρα δίνουμε το λόγο στους συντονιστές. Πρώτος, για το ΕΛΚΑ ο κύριος Καρλ Χάιντς. Και μετά είναι ο κύριος Γκουλάιν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, με πολύ χαρά άκουσα το φιλόδοξο πρόγραμμα, πρόγραμμά σας. Ειλικρινά μου, πρέπει να πω, ε, είστε για μένα η 46η Προεδρία και έχω ακούσει πολλές ε, ελπιδοφόρες διακηρύξεις που πάντα με εντυπωσίαζαν. Αλλά η Προεδρία του Συμβουλίου δεν έχει ως ρόλο μόνο να χειροκροτεί τις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της όταν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση από κοινού να εφαρμόσουν τις κοινέ ε, αποφάσεις. Αυτό είναι παλιό παραπονό μου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κι εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τις χώρες οι οποίοι αποφασίζουν από κοινού, οι οποίες αποφασίζουν εδώ και χρόνια από κοινού μέτρα τα οποία μετά δεν εφαρμόζουν. Ε, μιλήσατε για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την ε, πολιτική για τα απόβλητα. Είναι καταστροφή. Χάος κατά την εφαρμογή. Καμία προσπάθεια να βασιστούμε στα κοινά κριτήρια. Τι θα κάνετε σε σχέση με αυτό. Βεβαίω η Επιτροπή είναι θεματοφύλαξη των συνθήκων, αλλά είστε Προεδρεύων του Συμβουλίου. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε ευθύνη να εφαρμόσουμε αυτά που και τα τρία θεσμικά όργανα αποφάσισαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και από την πλευρά μας, καλώς ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Ο Ματίας Γκρότο, ο Πρόεδρός μας, ε, ήταν ενθουσιασμένος κατά την επίσκεψή του ε, για το Άτυπο Συμβούλιο Όλοι οι προεδρεύοντες έρχονται με θαυμάσιες προθέσεις, θαυμάσιους στόχους. Πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσετε να εφαρμόσουμε τουλάχιστον εν μέρη αυτούς τους στόχους. Χαιρετίζω αυτό που είπατε ότι πρέπει να είναι πρωτοπόρα Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σαφές, απτό θα έλεγα, ότι αναμένει ο κόσμος μια μεγάλη αλλαγή προς μια πράσινη οικονομία, προς ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης και η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη ευθύνη και από ιστορικής πλευράς. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε πότε θα αποφασίσουν όλοι να κάνουν κάτι. Πρέπει να προχωρήσουμε. Το μεγάλο θέμα στο Ρίο ήταν η βιωσιμότητα. Το 2001 είχαμε μια στρατηγική βιωσιμότητας είχε διατυπωθεί στο χαρτί. Ερώτηση προς εσάς, θα αναλάβετε μετά το Ρίο πρωτοβουλίες ούτως ώστε να αναβιώσει, να ξαναζωντανέψει η στρατηγική βιωσιμότητα. Έχει εξαφανιστεί. Έχει διάφορες επιγραφές, διάφορους τίτλους. Μιλάμε πάντα για οικονομική, κοινωνική, βιώσιμη κτλ. ανάπτυξη, αλλά στην πράξη έχουν εξαφανιστεί. Χαίρομαι που αναφερθήκατε για το 7ο πρόγραμμα για το περιβάλλον το έκτο αυτή τη στιγμή ακόμη τρέχει, αλλά υπάρχει ένα κενό μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται το έβδομο. Η Προεδρία σας θα μπορούσε να θέσει τους πρώτους στόχους. Πρώτα απ' όλα να μειωθεί ακριβώς αυτή η έλλειψη εφαρμογής των αποφασισμένων. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, όπως ανέφερε και ο Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Έχουμε πολλούς νόμους και δεν τους εφαρμόζουμε. Και επίσης, αυτή η προσπάθεια συλλογικής πρόθεσης όλων των στόχων να καταλήγει σε έναν κοινό παρανομαστή, δηλαδή την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό πρέπει είναι ο στόχο του 7ου προγράμματο για το περιβάλλον. Θα περιμένω λοιπόν ε, εναγωνίω τι προόδου. Τρίτον, είμαστε σε περίοδο οικονομική κρίση. Οπότε κινδυνεύει να εξαφανιστεί η περιβαλλοντική πολιτική. Μιλήσατε για το screening για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα επίση ε, να ζητήσω να υπάρξει και screening του προπολογισμού, Επανειλημμένα το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει και για τη δημοσιονομική πολιτική να κάνουμε προσπάθεια θεωρητική εξέταση πώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να παίξετε λοιπόν ρόλο σημαντικό γι' αυτό και για τον προπολογισμό του 2013 βεβαίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρο Τζο. Κρι Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα για την ανταλλαγή εκπομπών έχει δυσχέρειες αυτή τη στιγμή, για την εμπορία εκπομπών, συγγνώμη, έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός ε, εκπομπών για ε, ε, εμπορία και είναι πολύ χαμηλή τιμή. Οι εταιρείε ηλεκτρισμού παρακαλούν την Επιτροπή να διορθώσει την κατάσταση για να έχουν μια βεβαιότητα για τι επενδύσει πρέπει να κάνουν. Ξέρετε επίση ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο εάν ή όχι θα προωθήσει μια αναθεώρηση της αγοράς άνθρακα και να καθυστερήσει την ε, πώληση αδειών εμπορίας για να ανέβει η τιμή. Είπατε στις παρατηρήσεις σας ότι θέλετε να διατηρήσετε και να ενισχύσετε το σχέδιο εμπορίας εκπομπών ως Προεδρία καλείται την Επιτροπή να μας υποβάλει προτάσεις, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα αυτό είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του στην αντιμετώπιση των εκπομπών, που όλοι θα θέλαμε να παίξει. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για αυτά που είπατε για το εξάμεινο, όπως και οι συναδελφοί μου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας για τα θέματα αυτά και εγώ ως εισηγητής για τον κανονισμό εποπτείας φυσικά προσβλέπω στο να ολοκληρώσουμε την εργασία για το θέμα αυτό μαζί σας. Τρεις ερωτήσεις για θέματα που θα είναι πολύ σημαντικά το επόμενο εξάμεινο. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε λίγο περισσότερα για αυτά, θα ήθελα να μου πείτε. Πρώτον, κλιματική αλλαγή πώς θα αντιμετωπίσουμε στο εσωτερικό της Ένωσης. Ξέρουμε ότι έχει μπλοκάρει ένα κράτος μέλος το ε, ε, οδικό διάγραμμα για το, τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενώ τα άλλα 26 το υποστηρίζουν. Εάν περάσουν σε κανονισμό δεν υπάρχει πια βέτο. Ενώ αν είναι συμπεράσμα του Συμβουλίου και θέλουμε να εγκριθεί ένας οδικός χάρτης, τότε ακόμη και μία χώρα μπορεί να μπλοκάρει το θέμα αυτό. Τι προτίθεστε να κάνει το, προσεχές εξάμεινο για να αλλάξει η δική μας εσωτερική πολιτική. Για παράδειγμα, αν διαβάσουμε τον οδικό χάρτη που εγκρίνουν τα 26 κράτη-μέλη, καταλαβαίνουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να περάσουμε στο 25% το 2020. Διεθνώς επίσης, η κλιματική αλλαγή, η επιτυχία στην Τόχα είναι κλειδί για να συνεχιστεί το κιότο. Και ξέρουμε ότι οι κανόνες για να συνεχιστεί το πρωτόκολλο του Κιώτο είναι πολύ σημαντικοί. Και ένα από τα κουραστικά θέματα είναι τα AAUs, όπου μια συγκεκριμένη χώρα μπλοκάρει οποιαδήποτε συμφωνία. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, λύσει το πρόβλημα του AAU, δεν θα υπάρξει συνέχιση του Κιώτο. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό. Τρίτον, είστε και Υπουργό Γεωργίας. Αποφελούμε. Εδώ είμαστε Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ένα πολύ σημαντικό για την αναθεώρηση της ε, ΚΑΠ είναι το πρασίνισμα. Τι θα κάνετε ώστε το 30% της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ θα διατηρηθεί όταν θα συζητηθεί αυτή η τόσο ζωτική μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κιόλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Αν οι καλές προθέσεις ήταν ε, κριτήριο της, του αποτελέσματος, τότε σίγουρα θα επιτύχετε πολλά. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση ένα ειδικό θέμα που αφορά την Κύπρο. Ένα για το οποίο σας έγραψα προσωπικά. Αλλά θα ήθελα ε, να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την παράνομη παγίδευση πουλιών. Φαίνεται ότι ακόμη και 2, έως 2,8 εκατομμύρια πουλιών ε, πιάστηκαν σε παράνομες παγίδες. Και το φθινόπωρο είναι βέβαια η ακμή αυτής της περίοδου. Τι θα κάνει η Κυπριακή Προεδρία ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τζούλη. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Να δώσω και πάλι το λόγο σε εσάς κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές ε, παρεμβάσεις. Παρόλο που σέβομαι τον χρόνο όλο, θα είμαι σύντομος στις απαντήσεις μου για να δοθεί και ευκαιρία σε όλους που βάλουν και άλλες ερωτήσεις. Αναφορικά με την αηφόρο ανάπτυξη που λέχθηκε από αρκετούς κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι υπήρξε έντονη κριτική για τα αποτελέσματα της διάσκεψης ιστορίου αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Αρκεί να δούμε, κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνος χρειάστηκε και προσπάθεια τα 27 κράτη-μέλη να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και μια κοινή γραμμή. Σίγουρα επιθυμούσαμε η διάσκεψη να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανάληψη δράσης. Το τελικό αποτέλεσμα ομολογουμένως δεν είναι τόσο φιλόδοξο, αλλά έγινε αποδεκτό ως ένας καλός συμβιβασμός. Ικανοποιητικά θεωρούνται μεταξύ άλλων και η ενσωμάτωση των θεματικών στόχων, η αποδοχή της πράσινης οικονομίας, έστω και σαν εργαλείο ενεργοποίησης πόρων, η έναρξη διαβουλεύσεων για διάφορα θεσμικά πλούσια. Από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, δεν ικανοποιεί για παράδειγμα η μη συμφωνία σε ουσιαστική αναβάθμιση του προγράμματος περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ενώ η υιοθέτηση των στόχων εφόρου ανάπτυξης φαίνεται ότι θα αργήσει. Η Προεδρία θα ετοιμάσει συμπεράσματα Συμβουλίου στο Συμβούλιο του Οκτώβρη προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόθεση όσων τουλάχιστον συμφωνήθηκαν. Πιθανόν το, στο Συμβούλιο του Δεκέμβρη να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις. Στο διεθνές τώρα επίπεδο είναι μέλημά μας να, να προωθήσουμε τις διαδικασίες για τα θεσμικά πλαίσια περιβαλλοντικής διαχείρισης και εφόρου ανάπτυξης με στόχους τα μέσα ελοποίησης, την βιοπικιλότητα περιοχών πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας και τη λειτουργικότητα του πλαισίου για το προγράμματα εφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. Αναφέρθηκε, κύριε Πρόεδρε, στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας σε συνέχεια των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο του Ιούνιου η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει το θέμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό έχοντας προγραμματίσει τη συζήτησή του σε δύο συνεδρίες της Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος τον Δεκέμβριο προγραμματίζεται παρουσίαση του προγράμματος από την Επιτροπή σε περίπτωση όπως είπα που υπάρχει αντικείμενο θα ετοιμαστεί και μια έκθεση πρόοδου. Από τα συμπεράσματα όμως του Συμβουλίου τον Ιούνιο σημειώνεται το όραμα 2050 και η στόχη 2020 προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλύτερη επιβολή και ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάτι στο οποίο αναφέρθησαν αρκετοί ευρωβουλευτές, καθώς και οι τομείς των νερών, των αποβλήτων και προστασίας της φύσης, εμείς σαν Κυπριακή Προεδρία θεωρούμε ότι το πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου και τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Τέλος πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός διασύνδεσης με τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Ρίο, ώστε σχετικές δράσεις και στόχοι από αυτά να περιληφθούν και στο νέο πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα δράσης. Τώρα αναφέρθηκε, αναφερθήκατε στο θέμα του δρόμου για την Τόχα, για την κλιματική αλλαγή. Οι θέσεις μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσκεψη της Τόχα θα συμφωνηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος τον προσεχή Οκτώβρη όταν θα έχουμε και τα συμπεράσματα Συμβουλίου. Είναι επιθυμητή έκβαση στην Τόχα να είναι ένα αποτέλεσμα που θα περιλαμβάνει και την υιοθέτηση μιας δεύτερης περίοδου δεσμεύσεων από την 1η του Γενάρη 2013, να προωθηθούν οι διεργασίες για μια νέα νομικά δεσμευτική συμφωνία το αργότερο μέχρι το 2015, η οποία να ισχύει για όλα τα μέρη, να προωθηθεί το πρόγραμμα για να ενισχυθούν οι στόχοι μείωσης εκπομπών μέχρι το 2020 που αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια παγκόσμια προσπάθεια και να ενεργοποιηθεί το Πράσινο Ταμείο της Επιτροπής Προσαρμογής και του Μηχανισμού Τεχνολογίας. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για να γεφυρωθεί η ολοκλήρωση της περίοδου ταχείας εκκίνησης χρηματοδότησης το 2012 με την έναρξη της περίοδου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως 2020. Εμείς σαν Προεδρία θα συζητούμε τακτικά με τους έντιμους ευρωβουλευτές για την πρόοδο των εργασιών. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου θα τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και οι ευρωβουλευτές που θα είναι μαζί μας στην Τόχα σίγουρα θα έχουν μια ενεργό προσέγγιση σύμφωνα με τις θέσεις της Ένωσης οπότε ελπίζουμε στο καλύτερο. Αναφέρθηκε ο δικός χάρτης για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που είναι μια μεγάλη πρόκληση θα πρέπει να ομολογήσουμε ειδικά με την τωρινή οικονομική κατάσταση ως Κύπρος ε, συμμετείχαμε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης της πρότασης και υποστηρίξαμε τα σχετικά συμπεράσματα που προτάθηκαν για ταχεία περίοδο όσον αφορά τη στρατηγική για χαμηλές εκπομπές άνθρακα το 2050. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια αρνητική εξέλιξη στο φάκελο. Ε, καμιά αλλαγή έχει γίνει όσον αφορά τις θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τις οποίες κύριε Πρόεδρε δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και δεν έχουμε προγραμματίσει νέα πρωτοβουλία για το θέμα. Θα είμαστε όμως έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια στις συζητήσεις πολιτικού επίπεδου και να εξετάσουμε τρόπους για βήματα προς τα εμπρός σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. όσον αφορά τα θέματα των αποβλήτων υπάρχουν στις διάφορες νομοθεσίες και στους κανονισμούς αρκετοί όροι και πρόνοιες που η Επιτροπή πρέπει να επιτηρεί και να ελέγχει η ελοποίησή τους αφορούν όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εφαρμογή των όρων αυτών σε πρώτη ευθύνη και πρώτη προτεραιότητα και πολύ λιγότερο την Προεδρία παρόλο που θα συμβάλλουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Επειδή είμαι και Υπουργός Γεωργίας, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι για το θέμα του πρασινίσματος του πρώτου πυλώνα της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής και της κοινή αλληλευτικής πολιτικής γιατί μιλάμε και για τις δύο πολιτικές, εμείς ε, ως Κύπρος αντιμετωπίζουμε πολύ θετικά καταρχήν τις βασικές αρχές, πάνω στις οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και συμφωνούμε με την μεγιστοποίηση της συμβολής των γεωργών στην παραγωγή των δημόσιων αγαθών από τη μια, αλλά και με τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν οι γεωργοί μας για το πρασίνισμα της, Κυπρια... της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ε, επίσης, για το θέμα αναφέρθηκα στην κοινή αλλιευτική πολιτική. Συμφωνούμε με το πρασίνισμα με την έννοια της αλίευσης σε επίπεδα που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των αποθεμάτων και να προσφέρουν υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Αναφέρθηκε έγινε αναφορά για την παράνομη παγίδευση και θανάτωση των άγριο πτηνών, που η Κύπρος ε, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσει και, αν, τελικά να εξαλείψει την παράνομη παγίδευση των πτηνών. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Μεταξύ του 2001 και 2011 εντοπίστηκαν και καταγγέλθηκαν συνολικά 3.600 περιπτώσεις λαθροθυρίας, από τις οποίες οι 1.700 περίπου αφορούσαν παράνομη παγίδευση και σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούσαν παράνομο εμπόριο άγριων πτηνών σε εστιατόρια. Καταγγέλθησαν 25 ιδιοκτήτες εστιατορίων, ενώ ένας σημαντικός αριθμός εστιατορίων σταμάτησαν να διαθέτουν άγρια πτηνά διεξάγουμε πολύ συχνά εκστρατείες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμόρφωση με τις νομοθεσίες. Το ζήτημα αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το δικό μας κράτος. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την παράνομη θανάτωση των πτυνό που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2011 στη Λάρνακα αν και το φαινόμενο της παράνομης ε, παγίδευσης ψινών δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί, είναι τώρα πιο ελεγχόμενο και τα περιστατικά έχουν μειωθεί σημαντικά. Η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας και ευαισθητοποίηση του κοινού παραμένουν το κλειδί για την ουσιαστική λύση του προβλήματος. Αυτά σε γενικές γραμμές, κύριε Πρόεδρε. Ε, αν επιθυμείτε να συνεχίσουμε με, την, με τις ερωτήσεις, είμαι πρόθυμος να δεχτώ οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις τεθούν. Chairman, I wonder if the minister... Πρόεδρε, δεν ξέρω αν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή. Ρώτησα, ρώτησα συγκεκριμένα εάν η Προεδρία θα καλούσε την Επιτροπή να κάνει προτάσεις για να τεθούν κατά μέρο κάποιες άδειες, ούτως ώστε να ενισχυθεί, δηλαδή να μην πολυθούν τώρα οι άδειες για να ενισχυθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πρόεδρος, ωραία, θα είναι για το δεύτερο γύρο. Ας αρχίσουμε το κατάλογο των ομιλητών. Αρσένης, Εστρέλα και μετά θα δούμε. Α, και Μπράντι. Αλλά πρώτος ο κύριος Αρσένης. Πρόεδρε, Με... θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την, ε, και σας Υπουργέ και την ε, Κυπριακή Προεδρία για την οργάνωση, την ε, σοβαρότητα και τη φιλοδοξία της Προεδρίας σας και στα θέματα περιβάλλοντος. Είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση και της ατζέντα Προεδρίας στα θέματα υγείας χθε και χαιρόμαστε που συνεχίζει να είναι το ίδιο επίπεδο η παρουσία στα θέματα περιβάλλοντος. Ρώτησα τους πολίτες τι θέματα να σας, έθεσα, έθετα σε αυτή τη συναδρίαση και οι πολίτες βάλαν σε προτεραιότητα την ΚΑΠ. Ε, απαντήσατε βέβαια σε αυτό το ζήτημα, την, ε, ε, την πρωτοβουλία σας για την προστασία των εργαζομένων από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, αν θα είχατε τις πρωτοβουλίες, και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών δασών μέσω της χρήσης μη πυρόφιλων δέντρων όπως η πελανιδιά. Ήταν κάποια τα ερωτήματα. Θα ήθελα να σα θέσω όμως ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το Ρίο αναφερθήκατε στο τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε στο Ρίο. Και αληθεύει ότι η συμφωνία δεν ήταν στο επίπεδο της φιλοδοξίας που θα θέλαμε. Ε, όμως έχουμε μια δύναμη συμφωνία στα χέρια μας με, με ασαφή πολλές φορές ε, διατύπωση των δεσμεύσεων που έχουμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε πλήρω και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το αν θα είχαμε μια δυνατή συμφωνία που δεν θα, που δεν θα εφαρμόζαμε. Ε, έχετε το σκοπό ή σκοπεύετε να εξετάσετε τη δυνατότητα να αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την Προεδρία σας ε, την πρωτοβουλία να, να κινητοποιήσει τις διεθνείς εξελίξεις στα δύο θέματα που έχουμε αδύναμη φρασολογία που είναι το να κινηθούμε πέρα από το GDP, πέρα από το ΑΕΠ προς ένα νέο, ε, πιο, ένα νέο δίκτυ ε, ανθρώπινης ανάπτυξης αλλά και προς την δημιουργία πραγματικά του παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ για την τόσο σαφή σας παρουσίαση του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας. Μου άρεσε ιδιαίτερα η αποφασιστικότητα που επιδείξατε για την ευόδοση του έργου σας. Ο συνάδελφος Τζον Λάινεν αναφέρθηκε στο πόσο δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του Ρίο συν 20. Εμείς διαπιστώνουμε όμως και τα τελευταία χρόνια ότι όλες αυτές οι διεθνείς συναντήσεις δεν οδηγούν σε, στα ευελπιστούμενα αποτελέσματα. Η τελευταία διάσκεψη για το κλίμα δεν οδήγησαν σε αποτελέσματα. Αποτέλεσαν πραγματική πτώχευση. Το Ρίο συν δεν προσέγγισε καν τις προσδοκίες μας. Στο μεταξύ, οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα, η υπερθέρμαση του πλανήτη. Επίσης, η απερίμωση συνεχίζεται, οικοσυστήματα καταστρέφονται. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, και ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε μια νέα διάσκεψη αφιερωμένη στην βιοπικιλότητα. Ρωτώ, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για αυτή την εντέκατη διάσκεψη για την βιοπικιλότητα. Προβλέπετε ότι θα έχουμε σημαντικές πρόοδους έναντι της διάσκεψης της Ναγκόγια ή πάλι θα αναβάλουμε εσαΐ τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, Κέρτιν Γιάνν και Μπράντι, επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την διάσκεψη του ρίου. Βέβαια είμαστε απογοητευμένοι όλοι από την ε, κατάληξη, το τελικό κείμενο του Ρίο. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η πολυμερής ε, προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω δεν έχει τα αποτελέσματα που αναμέναμε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε την στρατηγική μας για να, επιδιώξουμε, για να επιτύχουμε την, το πρασίνισμα της παγκόσμιας οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν μια πολύ πιο πραγματιστική προσέγγιση. Να στοχεύσουμε περισσότερο άλλους τομείς πολιτικής. Ένας εκ των οποίων είναι ο τομέας της αναπτυξιακής πολιτικής και ο άλλος είναι η εμπορική πολιτική. Και για τους δύο τομείς αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ μεγάλος παράγων στην παγκόσμια σκηνή. Θα θέλατε να πάρετε πρωτοβουλία να πείσετε τους συναδέλφους σας ότι η αναπτυξιακή πολιτική και η εμπορική πολιτική θα μπορούσαν να λαμβάνουν πολύ περισσότερο στο εσωτερικό τους υπόψη την ε, περιβαλλοντική πολιτική, να χρησιμοποιούμε δηλαδή τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και την αναπτυξιακή μας πολιτική, ούτως ώστε να βοηθήσουμε άλλες χώρες να πρασινίσουν την οικονομία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννη. Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Η Προεδρία της Κύπρου έκανε καλή προπαρασκευή και ήδη στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις το Μάιο στη θαυμάσια χώρα σα διαπιστώσαμε ότι είχατε καλά προπαρασκευαστεί. Σήμερα όταν μιλήσατε για τη Γεωργία είπατε ότι υποστηρίζετε την κοινή γεωργική πολιτική στη βάση. Θεωρείτε ότι είναι καλό να υπάρχει το πρασίνισμα. Αλλά αν σκεφτώ το νησί αυτό Έχετε ένα θαυμάσια, μια θαυμάσια γεωρική παραγωγή, θαυμάσια φρούτα. Αλλά αυτά που είπατε για το οικολογικό δάσος, πώς θα το ορίσουμε. Τι θα συνέβη δηλαδή, ότι κάποια εδάφη που τώρα παράγουν θα βγουν από την παραγωγή και θα γίνουν χέρσα περιοχή. Δεν ξέρω εάν το κάνετε αυτό, αν συμφωνείτε με τον Επίτροπο. Δεν ξέρω αν είναι συνολικά η καλύτερη αντιμετώπιση και αν με αυτόν τον τρόπο προωθούμε αρκετά την οικολογική διάσταση. Θέλουμε να επιτύχουμε κάτι στο μέλλον. Η Προεδρία πρέπει να το συζητήσει αυτό μαζί μας. Αυτό ισχύει και στην συζήτηση που κάναμε και χθε για, τις, για τα σχέδια δράσης, για ε, τις εκπομπές ε, ε, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και για το πώς θα τις μειώσουμε σε σχέση και με την δασοκομική πολιτική κομισιόν συνδυάζει τη δασοκομεία με την πολιτική καλλιεργημένων γεών. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτή η συμπερίληψη και ο συνυπολογισμός οδηγεί σε πολλή γραφειοκρατία και στο τέλος θα έχουμε μηδέν κέρδος και για το περιβάλλον και για τη γεωργία. Αξίζει λοιπόν τον κόπο αυτή η προσέγγιση. Ή θα πρέπει να εξαγάγουμε τη Γεωργία από αυτήν την αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπελιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα φιλόδοξα σχέδια για το περιβάλλον κατά την ε, Κυπριακή Προεδρία. Εγώ, σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων, θα ήθελα να μπω σε όλη αυτή τη σειρά σκεπτικού για το αμέσως μετά το Ρίο, δηλαδή για την 11η συνδιάσκεψη για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Εσείς κάνατε την εξαγγελία και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα τρία κεφάλαια ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θα μεταφερθεί από το Συμβούλιο και το πώς θα οριστεί. Η, η συνέχεια Έχετε ένα νομοθετικό πακέτο με προθεσμίες. Θα επικυρώσετε το πρωτόκολλο της Ναγκόγια στους επόμενους έξι μήνες. Θα καλέσετε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να επικυρώσουν αυτό το πρωτόκολλο. Και όσον αφορά στη χρηματοδότηση, θα ξεκινήσετε τη συζήτηση για, τις, ε, για τους νέους πόρους, για τις νέες πηγές χρηματοδότησης και για το θέμα της αιρεσιμότητας ε, ε, των δημοσίων ενισχύσεων ε, κυρίως μέσα στα πλαίσια αυτών των δημοσίων ενισχύσεων στα πλαίσια της ΚΑΠ για την βιοπικιλότητα και εσείς είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε ένα φάκελο σχετικά και για το τελικό στρατηγικό σχέδιο Νταϊσί σχετικά δηλαδή με τις βλαμπερές επιπτώσεις ε, στη βιοπικιλότητα. Εσείς ε, τι θέλετε να κάνετε, πώς θα συνεχίσετε το ρίο για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους ωκεανούς και για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Θα ξεκινήσετε στο Συμβούλιο τη συζήτηση για μια οδηγία πλαίσιο για το έδαφος. η κυρία Κονή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ έχω δύο διαφορετικά θέματα που θέλω να θίξω. Το πρώτο αφορά στην πολιτική συνοχή, στην περιφερειακή πολιτική, για την οποία έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος και ήμουν εγώ η εισηγήτρια. Για αυτή τη γνωμοδότηση έλεγα ότι η πολιτική στον τομέα αυτό λαμβάνει υπόψη της την υποδομή για το νερό αλλά και για την εξυγίανση της υποδομής υδροδότησης κυρίως στις χώρες όπου είναι παλιές οι εγκαταστάσεις. Ας πούμε στη Γαλλία το νερό το οποίο μαζεύεται στα φρεάτια μέχρι να φτάσει στα νοικοκυριά ε, χάνεται το 40% και αυτό λόγω της αρχαιότητας της υποδομής. Είναι δύσκολο λοιπόν για, τους, ε, για τη δημόσια, για την, συγγνώμη, την τοπική αυτοδίκηση να αναλάβει την εξυγίανση αυτού του δικτύου. Ρωτώ λοιπόν μέσω του Φεντέρ μήπως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε ένα μέρος αυτής της επισκευής. Τώρα, για την ηλεκτροκινητικότητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι που λειτουργεί πολύ καλά στις πόλεις, αλλά δεν το πολύ συζητάμε. Τι γίνεται όμως με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να, έχουμε, να, ε, ε, κάνουμε μεγάλες αποστάσεις. Πώς θα προβλέψουμε εμείς φορτωτές για αυτές τις μπαταρίες στις μεγάλες αποστάσεις και για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα ε, μηχανισμού φόρτισης των μπαταριών χρειάζεται χρηματοδότηση σε αυτά τα σημεία κινητικότητας. Ε, χρειάζομαι υποστήριξη της Προεδρίας, διότι δεν είμαι σίγουρη ότι τα κράτη ε, θέλγονται από τέτοιου είδους σχέδια συγχρηματοδότησης είναι ένα σχέδιο το οποίο ε, θα, ε, θα ψηφιστεί αύριο στην ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, θα περάσει και από το Συμβούλιο αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, υποδομή για το νερό και η κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για μας. Τελευταίο σημείο για την πολιτική συνοχής, και το δέχτηκαν οι εισηγητές στην Ρέγγι, Ό,τι αφορά στα αθλητικά είδη και αυτά να χρηματοδοτούνται από την Κομισιόν, διότι είναι θέμα δημόσιας υγείας και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό. Τώρα, για το δικαίωμα φύτευσης αμπελιών. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα τα αμπέλια υπόκεινται σε ποσόστοση, σε δικαίωματα ε, φυτεύσεως. Εμείς στα πλαίσια της ΚΑΠ καταργήσαμε τις ποσοστώσεις και αυτό θα αρχίσει να ισχύει από το 2015 και μετά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την οικονομία του κρασιού, διότι αυτό το οποίο είναι η ουσία δηλαδή της ε, ε η, του οικονομικού συστήματος, ε, του κυκλώματος συγγνώμη, του κρασιού είναι η κατανάλωση και οι ποσότητες. Είδαμε τι απέγινε με την απολευθέρωση ορισμένων ε, προϊόντων όπως το γάλα που πραγματικά καταράκωσε όλο το δίκτυο του γάλακτος. Και η Κύπρος είναι μια χώρα που δεν υπέγραψε ή δεν υπέγραψε ακόμα αυτήν την ιδέα του να κάνουμε πίσω σε αυτό το δικαίωμα, στην άρση δηλαδή των, της ποσόστοσης ε, για τα αμπέλια. Λοιπόν, έχετε, ποιες είναι οι προθέσεις σας. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε την γνώμη σας και να δούμε την υπογραφή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα με ξέπετε αν δεν έπαιρνε το λόγο ο κύριος Ρίχα Τζέμπερ, που είναι ο συγκεκριτής για την έκθεση Blueprint. Οπότε, ε, τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο κύριος Ζέμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να κάνω μία ερώτηση για τα ύδατα. Κύριε Υπουργέ, έχω στενή επαφή με τους συνεργάτες σας για την πρόταση αυτή της Κομισιόν για τις κατά προτεραιότητα ουσίες στο νερό. Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο το θέμα αυτό ε, αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά από διάφορες χώρες. Ξέρουμε ότι μέσω της οδηγίας πλαίσιο είναι καλό, είναι αναυποχρεωμένη να υπάρξει συμφωνία μέχρι το 2015 και η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τακτικά ποιες ουσίες είναι σε αυτό το κατάλογο. Η πρόταση λοιπόν είναι ε, ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από ορισμένες χώρες μέλη όσον αφορά την συμπερίληψη φαρμάκων ή και κάποιων φυσικών ορμονών. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ακούσω την άποψή σας. Σε τι βαθμό δηλαδή είστε διατεθειμένοι να οδεύσετε και σε τι βαθμό θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστική η επίτευξη συμβασμών. Τι μπορείτε να κάνετε, για να το πω έτσι, να, τους, ε, να πείσετε κάποια κράτη-μέλη να σταματήσουν ε, τις προθέσεις τους σε σχέση με τις φαρμακευτικές ουσίες γιατί είναι σαφής κατάσταση όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων. Το επιχείρημα που αναφέρεται είναι βεβαίως σε μεγάλο βαθμό σωστό. Υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα υπέρ μιας τέτοιας ε, πρότασης, αλλά θα ήθελα να μάθω ποια είναι η πρόθεσή σας να κάνετε αυτή την ε, αναγκαία εργασία για να πείσετε ή εάν συμφωνείτε ότι αυτές οι τρεις ουσίες δεν θα έπρεπε να είναι στο κατάλογο του κατάπληκτου ουσιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. Έλεξε ο δεύτερος γύρος. Μία ερώτηση έχει μείνει επίση από τον πρώτο γύρο και κατόπιν η απαντήση από το δεύτερο γύρο. Κύριε Υπουργέ, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Πρόεδρε, ναι πράγματι έχει μείνει αναπάντητη η ερώτηση του κύριου Ντέιβις όσον αφορά τα AAUs Συμφωνώ ότι υπάρχει ακόμη πρόβλημα με τα EAUs. Κάποιες χώρες τα βλέπουν σαν assets, σαν ε, κάτι χρήσιμο και πολύτιμο. Αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία και πολύ σύντομα μάλιστα. Αναμένουμε την πρόταση της Επιτροπής για να προχωρήσουμε και με τις δικές μας πρωτοβουλίες αλλά όπως ανάφερα και στην ομιλία μου θα πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε το σύστημα των ATS με κάθε, με κάθε τρόπο. Δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω τόσο γρήγορα. Τώρα αναφερθήκατε για το Ρίο. Απλώς να πω ότι αρχίσαμε σήμερα στην ομάδα εργασίας για το περιβάλλον την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για το Ρίο και αναμένουμε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Θα δώσουμε σίγουρα κάθε προτεραιότητα στα δύο θέματα που ανάφερε ο κύριος Αρσένης, δηλαδή στις συμπληρωματικούς δείχτες και στο διεθνές πλαίσιο, για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά την στρατηγική για την βιολογική ποικιλότητα, εμείς ε, σαν Κυπριακή Προεδρία θα υποστηρίξουμε, όπως ανάφερα, τις παγκόσμιες αλλά και τις ευρωπαϊκές προσπάθειες που γίνονται για ανάσχεση της απώλειας της βιολογικής επικοινότητας. Είναι γνωστό ότι η επερχόμενη διάσκεψη στην Ινδία θα επιληφθεί αυτών των θεμάτων αλλά και θεμάτων κινητοποίησης πόρων. Έχουν τεθεί στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 που είναι όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να αποκατασταθεί η φύση. Ένα στόχος που είναι πραγματικά μεγάλο επίβολος. Εμείς ως Κύπρος φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ε, η νέα πρωτοβουλία για εξειδίκευση της χρηματοδότησης, γιατί ξέρετε καταλήγουν όλα τελικά στη χρηματοδότηση. Εδώ είναι που κολλούμε και πρέπει να το ομολογήσουμε ότι όταν είπατε ότι γίνονται διεθνείς διασκέψεις και δεν έχουν αποτέλεσμα, ξέρετε πολύ καλά ότι πίσω από αυτές τις, δεν θα τις πω αποτυχίες, αλλά τις, ε, τα μειωμένα αποτελέσματα, βρίσκεται η έλλειψη χρηματοδότησης. Η νέα πρωτοβουλία για εξειδίκευση της χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος LIFE υποστηρίζεται πλήρως από την Κυπριακή Προεδρία. Φυσικά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες για την βιοπικιλότητα και για το φύση 2000. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ότι στηρίζουμε τη χρηματοδότηση μέσω της κοινή αγροτικής πολιτικής. Το πρασίνισμα δηλαδή της γεωργίας και θεωρούμε ότι αυτό είναι πρωταρχικής ε, σημασίας και επειδή αναφέρθηκα και στην Αλία, ναι, πιστεύουμε ότι μέσα από το νέο Ταμείο Αλίας θα έχουμε δυνατότητες για προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των, των ειδών. αναφερθήκατε στις ουσίες προτεραιότητας για τα νερά. Ε, θα εργαστούμε για συμφωνία με τον κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας στα νερά. Αρχική επιδίωξη είναι η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφού πραγματικά το συντομότερο που θα επέρθει αυτή η συμφωνία είναι προς το, προς το συμφέρον όλων για να ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων των νερών. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εξέτασης του θέματος που μας έδωσε, κύριε Πρόεδρε, έτσι, λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες και απαραίτητες τροποποίησεις προκειμένου να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις στα πλέον δύσκολα θέματα. Λύσεις που μπορούν να γίνουν αποδεκτές και από τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών και από το Ευρωκοινοβούλιο. Χωρίς ε, να ξεχνάμε ότι πρέπει αυτές οι λύσεις να διασφαλίζουν και την προστασία του περιβάλλοντος. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θέματα στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφορούνται σε φαρμακευτικές ουσίες στον κατάλογο προτεραιότητας υποεπιτήρηση αλλά κάτι άλλο που ανησυχεί τα κράτη-μέλη είναι και το κόστος παρακολούθησης. Δεν πρέπει αυτό να είναι υπέρμετρα μεγάλο. Εάν παρόλες τις προσπάθειες δεν καταστεί δυνατή πίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο, που δεν το απέφχομαι, τότε θα επιδιώξουμε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο του, του Δεκέμβρη. Ε, έγινε αναφορά κύριε Πρόεδρε στην πράσινη ανάπτυξη που για μας η πράσινη οικονομία αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ανάπτυξη και πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίζεται ισότιμα σε όλες τις διαστάσεις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Φυσικά η μετάβαση στην πράσινη οικονομία προϋποθέτει και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών. Πρέπει να καταφέρουμε, κύριε Πρόεδρε, να εμβολιάσουμε και άλλες πολιτικές με πρασίνισμα και μιλώ φυσικά για πολιτικές ενέργειας, μεταφορές, βιομηχανία, πρώτες ύλες, γεωργία, αλία, Αλλά αν δεν αλλάξει πραγματικά η ανθρώπινη συμπεριφορά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Με την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τα αίτια που δημιουργεί η απουσία της πράσινης ανάπτυξης. Επειδή αναφέρθηκε για την χρηματοδότηση που απαιτείται για τη αλλαγή των υποδομών, για τα νερά, για τα δίχτυα που αναφέρατε της Γαλλίας που είναι πεπαλαιωμένα ή για την χρηματοδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να πω ότι ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχόλησε στο άτυπο συμβούλιο το περασμένο Σαββατοκυριακό ήταν η χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τέτοιες δράσεις, αλλαγή των δικτύων τοπορμήθειας για να μειώσουμε τις απώλειες ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα θεωρούμε ότι είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και είδαμε τρόπους που μπορεί να γίνει χρηματοδότηση. Δεν μπορεί πλέον να περιμένουμε όλα να τα κάνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός κάθε κράτους. Πρέπει να υπάρξει εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να υπάρξει συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, πρέπει να μπουν μέσα και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και ο ασφαλιστικός τομέας. Δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω όσες περισσότερες ερωτήσεις σημείωσα. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι οι ερωτήσεις τους έχουν μείνει πίσω, δεν είναι επίτητες που το έκανα, αλλά ε, μπορώ να συνεχίσω αν επιθυμείτε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ε, απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Είναι πλάτη πεδίο αρμοδιοτήτων. Μ' αρέσει η οριζόντια προσέγγιση που υιοθετείτε για βεβαίω την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγή σε συνδυασμό με την πολιτική υδάτων. Δεν είναι μεμονωμένα δηλαδή αυτά τα θέματα. Οι πολιτικές αυτές συνδυάζονται. Και επίσης αυτά που είπατε για τις διασκέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πώς στο μέλλον τώρα θα εκπληρώσουμε τα διεθνή καθήκοντά μας, πρέπει να το καθορίσουμε και ως Επιτροπή. Υπάρχουν μεγάλες ε, προσδοκίες ε, ενώπιον αυτών των ε, συνδιασκέψεων, αλλά να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να καθορίσουμε πρώτα απ' όλα τη θέση μας. Δηλαδή, Ίσως δεν θα σκόπουμε να την πούμε περιβαλλοντική ε, ε, συνδιάσκεψη, αλλά να την πούμε συνδιάσκεψη για ε, την αηφόρο ανάπτυξη. Άλλες περιοχές του κόσμου στοχεύουν περισσότερο στην κοινωνική διάσταση. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευαισθησίες των μεν και των δε, τις ευαισθησίες δηλαδή των εταίρων μας στο διεθνές επίπεδο. Είπατε πως δεν θα είσαστε ουδέτερος, μα φυσικά ως προεδρεύον δεν μπορείτε να είστε ουδέτερος. Και φυσικά αυτό δεν είναι πάντα ευχάριστο μόνο. Στην αρχή είναι πάντα ευχάριστη μια Προεδρία, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι πολλές φορές μιλήσαμε για τη συμφωνία για τις πρώτες αναγνώσεις. Καμιά φορά υπάρχουν αντιρρήσεις, ορισμένα θέματα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο. Γιατί το θέμα είναι η ποιότητα, όχι η ταχύτητα. Εμείς ως Κοινοβούλιο πηγαίνουμε σαν τρένο υψηλής ταχύτητας. Ε, περνάμε τα νομοθετήματα σαν τεζεβέ. Καμιά φορά όμως το Συμβούλιο είναι σαν ε, ατμομηχανή. Πηγαίνει πολύ αργά. Είμαστε γρήγοροι στο Κοινοβούλιο. Αλλά πολλές φορές ε, δεν πάνε όλα τα πράγματα τόσο γρήγορα. Σας παρακαλώ και το εξάμεινο και μετά το εξάμεινο ε, να λάβετε υπόψη και την αρμοδιότητά σας ως Υπουργός Περιβάλλοντος αλλά και ως Υπουργός Γεωργίας. Όταν είστε στο Συμβούλιο Γεωργίας να σκέφτεστε το πρασίνισμα της ε, πολιτικής γεωργίας και πείτε και στους υπουργού Οικονομικών ότι ε, θέλει παραδάκι αυτή η διαδικασία. Μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε μόνο εάν μετά δεν τα διαγράφουν όλα, δεν τα περικόπτουν όλα και μα αφήνουν ένα ελάχιστο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η πολιτική μα. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει. Οπότε για μας είναι πλεονέκτημα ότι συνδυάζεται αυτές τις δύο αρμοδιότητες. Σας παρακαλούμε, κέντρο της προσοχής σας να είναι πάντα η περιβαλλοντική πολιτική και είπατε ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι το αποφασιστικό. Είναι όπως είναι, εδώ πρέπει ορισμένες φορές και τα τρία θεσμικά όργανα να κάνουν καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Γιατί θέλουμε κάτι να αντιμετωπίσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καμιά φορά δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρούμε στο μέλλον το χρόνο για να συζητάμε με τους ανθρώπους, γιατί μόνο τότε μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ατόμων. Σας εύχομαι καλή δύναμη, αντοχή και κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Πρέπει να πω ότι ό,τι έχω δει μέχρι στιγμή έχετε πολύ καλά προετοιμαστεί, αλλά ένα είναι σίγουρο. Όπω πολλέ προεδρίε που είχαν προετοιμαστεί καλά, στο τέλο θα ε, κριθείτε με βάση τα αποτελέσματά σα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι μια ομάδα. Πρέπει λοιπόν η ομάδα να έχει καλή απόδοση συνολικά. Ξέρω ότι έχετε προετοιμαστεί καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σα εύχομαι πολύ πολύ επιτυχία. Ε, απλώς κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξαναναφέρω ότι τον Νοέμβριο με το συνέδριο μας στην Κύπρο για το Blueprint και θα ήταν ιδιαίτερη μας τιμή εσείς αλλά και άλλοι έντιμοι ευρωβουλευτές εάν μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Και επίση είναι αυτονόητο κύριε Πρόεδρε ότι οποτεδήποτε χρειαστεί να παρευρεθώ στην Επιτροπή σας. Είμαι πρόθυμος να το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπαμε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και θα κρυθείτε από τα αποτελέσματα. Οπότε, μετά την παρουσίαση της Προεδρίας, να συνεχίσουμε με τις δικές μας δραστηριότητε. Συγκεκριμένα νομοθετήματα, λοιπόν. 16. Ασφάλεια των δραστηριοτήτων γεώτρησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοιχτής θαλάσσης όπως μπορείτε να καταλάβετε είναι ένας πολύ σύντομος αλλά πολύ σημαντικός τίτλος Ίσως δεν είναι ο πιο κατάλληλος παρόλα αυτά αλλά θέλουμε να υπάρξει ε, σαφήνεια Οπότε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση Α, Κρήτον. Ο Κρήτον αντικαθιστά τον εισηγητή. Παρακαλώ, Κρήτον. Thank you very much. Uh, I will be... Ευχαριστώ. Θα διαβάσω τις παρατηρήσεις του κυρίου Παλέτσκης, ο οποίος δεν μπορούσε να παρευρεθεί, δυστυχώς. Οι σύγχρονες κοινωνίες ζητάνε από τις εταιρείες να βρουν καινούρια παιδεία και καινούριε τεχνικέ για να μπορούν να εξορίξουν όλο και βαθύτερα στι ανοιχτέ θάλασσε. Αλλά επειδή λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και εξοικονομήσεις, οδηγεί στο να μην λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια. Μπορεί να έχει επίση ε, βλαβερέ, καταστροφικέ επιπτώσει στο περιβάλλον όπω έγινε τον τύπο του Horizon στο κόλπο του Μεξικού πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Και κατόπιν ο κύριο Παλέτσκης καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν, θεωρεί το κατάλληλο μέσο για να υπάρξει αναγκαία ασφάλεια και περιβαλλοντικά στάνταρ παντού στην Ένωση. Ωστόσο, όπως αναφέρει, είναι πεπισμένος ότι θα υπάρξουν μια σειρά τροπολογίες που θα ενισχύσουν την πρόταση, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματική. Το πιο επίμαχο θέμα είναι ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Εκπρόσωποι του κλάδου και διάφορα κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερη μια οδηγία. Σημειώνει ο κύριος Παλέτσκης ότι σε προηγούμενες συζητήσεις στην Ήτρε 90% της συζήτησης έγινε γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Κατά τη γνώμη του κύριου Παλέτσκης και η γνώμη των σοσιαλιστών είναι, είναι να υποστηρίξουν την θέση της Κομισιόν θεωρώντας ότι ένας κανονισμός θα βοηθούσε να υπάρξει θεμητός ανταγωνισμός παντού στην Ένωση. Ούτως ή άλλως πρέπει το νομοθέτημα να είναι εφαρμόσιμο για να διασφαλίσουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια και των πολιτών και του θαλάσσου περιβάλλοντος διασφαλίζεται κατά το μέγιστο κατά τις ενέργειες εξόρυξης στα ανοιχτή θάλασσα. Οι εταιρείε θα έπρεπε να έχουν ε, δεσμεύσει επαρκείς πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, ένα μεγάλο δυστύχημα της επιπτώσεις τους και το καθάρισμα της περιοχής. Αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της ε, κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής ο Μολύνων πληρώνει. Εάν γίνουν μεγάλα ατυχήματα, πολλές μεγάλες εταιρείες, αλλά ακόμη περισσότερο οι μικρές μπορεί να πτωχεύσουν. Οπότε θα αναλάβουν φορολογούμενοι. Αυτές οι οικονομικές λοιπόν πρέπει να εξαρτώνται από το βαθμό ανάληψης κινδύνων σε τέτοιους χώρους εξόρυξης στην ανοιχτή θάλασσα. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε την ενημέρωση του κοινού με βάση την διεθνή νομοθεσία. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης έγκαιρα για το ενδεχόμενο Εξερεύνηση και εξόρυξης στην ανοιχτή θάλασσα. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τα μεγάλη κλίμακας ατυχήματα και πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο για να περιοριστούν οι ζημίες και στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Επίσης πρέπει όσοι κάνουν καταγγελίες ανώνυμα πρέπει να προστατεύονται. Οι αρχές που χορηγούν άδειε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα ευαίσθητα ε, θαλάσσια οικοσυστήματα όταν χορηγούν τέτοιες άδειε εξόρυξης. Προτεραιότητά μας δεν θα πρέπει να είναι το βράχυπρόθεσμο οικονομικό κέρδος, αλλά η μακροπρόθεσμη βιώσιμη εξόριξη. Οι εταιρείε πρέπει να έχουν σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών που να ελέγχονται τακτικά για να είμαστε σίγουροι ότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός είναι καταλήλου επίπεδου. Το επίπεδο αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό ακόμη όταν λειτουργούν και εκτός των ορίων της Ένωσης. Πρέπει να πείσουμε τις μη κοινοτικέ χώρες, ιδιαίτερα όσες έχουν τέτοιου τύπου δραστηριότητες κοντά στα σύνορά μας, να εγκαθιδρύσουν τέτοιες προβλέψεις. Διάφορες γειτονικέ μας χώρες θα πρέπει να κάνουν από κοινού με τις ε, δικές μας ε, υπηρεσίες επιθεωρήσεις. Σωστή ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ προστασία του περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας από τη μια μεριά και των συμφερόντων των εταιριών για να βρούμε νέους ενεργειακού πόρους. Εάν υπάρξουν μεγάλης κλίμακας ατυχήματα, πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά σχέδια ανταπόκρισης και αντίδρασης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια αυτά είναι παντού στα ύδατά μας προς εφαρμογή. Είτε είναι κοντά στις ακτές, είτε σε πιο επικίνδυνες περιοχές όπως η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα. Ένα τέτοιο κείμενο θα πρέπει να είναι ένα τεστ αντοχής για όλες τις δραστηριότητε παντού στα ύδατά μας για να διαπιστώσουμε πού είναι οι πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις και να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει με την υγεία των πολιτών διασφαλίζοντας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στην ε, σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω τώρα. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Παλέτσκης, αλλά φυσικά και τον κύριο Αρσένη που μας παρουσίασε το θέμα αυτό σήμερα. Ευχαριστώ για το σχέδιο. Καλωσορίζω τις προτάσεις της Κομισιόν που τονίζει την ασφάλεια τέτοιων δραστηριοτήτων ανοιχτής θαλάσσης, αυξάνει την ασφάλεια μάλιστα και προσπαθεί να μειώσει τις επιπτώσεις των ατυχημάτων. Η πρόταση αυτή για μένα που είμαι από τη Βόρεια Γερμανία, αλλά και από άλλους που ζουν σε παράκτες περιοχές, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ξέρουμε όλοι τι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον έχουν τέτοιου τύπου ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου χίλιες τέτοιες εγκαταστάσεις ανοιχτής θαλάσσης. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο μέλλον θα είναι περισσότερες. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις εξόρυξης βεβαίως δημιουργούν ένα συγκεκριμένο μάλιστα μεγάλο κίνδυνο. Όπως τον περιέγραψε ο κύριο Αρσένης, είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο να ενοποιηθεί, να υπάρχει ένας κανονισμός. Θα ήταν το ελάχιστο να καθορίζει λοιπόν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Για την πρόταση του κύριου Παλέτσκης θέλω να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, η συγκεκριμένη αλλαγή για να αυξηθεί η διαφάνεια. Πολύ καλή. Δεύτερον, χαιρετίζω τη συμπερίληψη για την διάλυση των εγκαταστάσεων. Φυσικά πρέπει από τώρα να διασφαλίσουμε ότι όταν στο μέλλον οι δραστηριότητε μια εγκατάσταση λήγουν, θα είναι εγγυημένη ασφάλεια κατά την ε, αποσυναρμολόγησή τη. και συγκεκριμένα το κράτο μέλο όπου γίνονται αυτέ τι εργασίε πρέπει να έχει δυνατότητα να ζητήσει να γίνουν κοινέ επιθεωρήσεις. Η όλη αυτή η διαδικασία βεβαίω μπορεί να κρατήσει πολύ και αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Με κοινούς κανόνες είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και δεν χρειάζονται πολύ περαιτέρω, ε, πολλές περισσότερες διατάξεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άχιατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κρήτονα που έκανες αυτήν ε, την δουλειά Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την γνωμοδότηση. Σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζουμε την κατεύθυνση του κυρίου Παλέκη, τον προσανατολισμό του. Υποστηρίζουμε λοιπόν τον εισήγητη και νομίζω ότι καλό να ενδυναμώνουμε τις προτάσεις της Επιτροπής, διότι ήταν κάπως απογοητευτικές και πρέπει να πω όταν δημοσίευσαν ε, τις προτάσεις πέρσι, μας απογοήτευσαν κάπως. Νομίζουμε ότι θα πρέπει συμφωνούμε ότι, ότι θα πρέπει να πρόκειται για κανονισμό και όχι για οδηγία. Υπάρχει κάποια συζήτηση κάπου ε, και υπήρξε κάποτε. Είναι καλύτερο να έχουμε έναν κανονισμό για να, ε, να μπορέσουμε να έχουμε ίσους όρους, να μην έχουμε μια συζήτηση για οδηγία ποιος θα εφαρμόζει τι ε, και να μην... και να μην επιβραβεύονται αυτοί που θέλουν να έχουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή ότι πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό. Η βασική ε, προτεραιότητα για κάθε γεώτρηση είναι να προλάβει ε, κάποιο, ε, κάποιο, ατύχημα σαν τον τύπο Horizon και θα πρέπει να χρειαστούμε επίσης μια επιθεώρηση των επιθεωρητών και ο ρόλος της ΕΜΣΑ είναι λογικό να υπάρξει μέσα στο πλαίσιο αυτό και αυτό λείπει από την ε, πρόταση της Κομισιόν αλλά και ο εισηγητής δεν αναφέρεται στην ΕΜΣΑ. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα ρόλο ε, στην υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας ε, την ευρωπαϊκή, διότι θέλουμε κάποια παρακολούθηση και εποπτεία στον τομέα αυτό. Όταν θέλουμε να προλάβουμε ατυχήματα θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ε, στις ευάλωτες περιοχές, στα ευάλωτα σημεία σε σχέση με τα οικοσυστήματα και σε σχέση με τις γεωτρήσεις που γίνονται σε μεγάλο βάθος θαλάσσιο. Αναφερόμαστε στην περιοχή του Βόρειου Αρκτικού, ωκεανού της Βόρειας Αρκτικής, όπου εκεί χρειαζόμαστε περισσότερη παρακολούθηση και χρειαζόμαστε τροπολογίες εφόσον υπάρξει πρόβλημα σε ατυχή κατάσταση, τότε ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η υπευθυνότητα. Ποιο είναι υπεύθυνο και εκεί συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, τι διατάξει, τα μέτρα, τα χρηματοδοτικά. Ε, θα πρέπει να ενισχυθούν, διότι είναι ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό το στάδιο ότι είναι οι ασφαλιστικέ εταιρείε ε, οι οποίε μπορεί να επισκέφθηκαν τα γραφεία σα επίση που λένε ότι δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε κατά το μάλλον ή τον Αυτό δείχνει πόσο το θέμα αυτό ενέχει κινδύνους. Ακόμα και οι ασφαλιστικές εταιρείε λένε ότι δεν ξέρουμε μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να ασφαλίσουμε διότι δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Και αυτό δείχνει ότι οι ε, πετρελαϊκές εταιρείες έχουν δραστηριότητες των οποίων οι κίνδυνοι είναι άγνωστοι. Και ποιος θα φέρει την ε, ευθύνη ε, τότε είναι το κοινό και όχι ο ιδιωτικός τομέας. Είναι ένα θέμα ο κίνδυνος αυτός που πρέπει να εξετάσουμε αν δεν μπορεί να ασφαλιστεί ε, από τι ασφαλιστικές εταιρείε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίες αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αυτής της δραστηριότητα και οι οποίες επίσης ε, εισπράττουν ε, τα κέρδη όπως η Shell α πούμε ότι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όχι δεν είναι ότι δεν πρέπει να είναι υπεύθυνε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να δεχθούμε την έλλειψη υπευθυνότητα τους, ούτε, όχι στα υδατά μας, ούτε στα υδατά μας, ούτε και εκτός ευρωπαϊκών υδάτων, όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείε ενεργοποιούνται και έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για ευρωπαϊκές εταιρείε, ακόμη και αν δρούν εκτός των υδάτων μας. Επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βεβαιωθούμε ότι θα είναι υπεύθυνε για το πλήρε κόστο και ακόμα και για την διάλυση, ε, απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών στο τέλο, ε, διότι αυτή η διάλυση επίση καλύπτεται από έξοδα των δημοσίων αρχών τελικό. Θα πρέπει λοιπόν αυτέ οι εταιρείε να παίρνουν τα κέρδη από τι δραστηριότητε, αλλά επίση να είναι και υπεύθυνε για όλη την αλυσίδα και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα το τονίσουμε αυτό στις τροπολογίες μας. Γενικά, υποστήριξη για τον προσανατολισμό ε, του εισηγητή για ενίσχυση του ρόλου της Κομισιόν, αλλά θα ε, προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ, Μπασάχιον. Και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο και Μπράντι, που εκπροσωπεί σήμερα το, την κυρία Λεπά. Σήμερα είναι η μέρα των αντικαταστατών, των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ, δεν μπορείς να έρθει η κυρία Λουπάζου Λίγες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον Κρήτονα και τον εισηγητή. Το σχέδιο γνωμοδότησης είναι πάνω από καλή αρχή. Θα υποβάλουμε ως φιλελεύθεροι κάποιες ευρωπολογίες για να ενισχύσουμε την έκθεση ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομικής, ε, των οικονομικών εγγύσεων και την ε, ανεξαρτησία των ε, ελεκτών. Χαιρόμαστε που δεν αλλάζει τη νομική βάση ο κύριος Παλέτσκης, το νομικό μέσον μάλλον. Ε, χαιρόμαστε που εμένει σε κανονισμό. Πολύ βασικός επίσης ο ρόλος της EMSA. Τώρα περιορίζεται στις μεταφορές ο ρόλος της. Η ομάδα μας θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να επεκταθεί ο ρόλος του οργανισμού αυτού για τη θαλάσσια ασφάλεια και στην εξόριξη και εξερεύνηση. Τώρα το θέμα της ε, υπετιότητας και της οικονομικής ασφάλειας αναφέρθηκε ήδη. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα ότι η Κομισιόν διευρύνει το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. Οι εταιρείε θα πρέπει κατά, τα κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής αυτών των εγκαταστάσεων να αποδεικνύουν ότι έχουν το επαρκές οικονομικό δυναμικό για να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές τους. Τέλος, Πρόεδρε. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανεξαρτησία των ελεκτών, των ανεξαρτήτων ελεκτών και η διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Μας ικανοποιεί ότι ο εισηγητής εισάγει την έννοια ε, ακραίων καταστάσεων Τώρα που ξεκινάμε, αυτό που ξεκινάμε σε αυτή τη φάση, εξόριξη στην Αρκτική. Πρόεδρος. Το λόγο έχει η Μαρίνα Γιάννη Κανάρκης που εκπροσωπεί τον συνάδελφο Στίβενσον. Ευχαριστή. Ναι, σήμερα είμαι Στίβενσον. Ναι, ναι, βελτιώνονται τα πράγματα. Θα διαβάσω από τις σημειώσεις του. Πρώτα απ' όλα Έχουμε όλοι πλήρη συνείδηση στο Κοινοβούλιο ότι η εξόριξη στην ανοιχτή θάλασσα περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους. Όπως ο συνάδελφος, η συνάδελφος είπε πέρσι, κάθε νομοθεσία για δραστηριότητες σε ανοιχτή θάλασσα θα πρέπει να εστιάζονται στο να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες να έχουν το υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να ε, μεριμνήσουμε, να μην υπερβάλλουμε τα πράγματα και υπάρχουν φόβοι. Η πρόταση αυτή ε, να θίξει την ενεργειακή ασφάλεια, ε, βγάζοντας ορισμένες εταιρείες από την αγορά από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαι υπερήφανος ε, για το ρυθμιστικό πλαίσιο στη Βόρεια Θάλασσα που είναι ένα παράδειγμα παγκόσμιο βέλτιστης πρακτικής ε, και χαιρετίζουμε ε, μερικά ότι μέρος του κειμένου της Κομισιόν βασίζεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι καλό, αλλά κράτη-μέλη να εξυψώσουν τα, τα πρότυπά τους και να έχουν υψηλότερο επίπεδο. Επίσης ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει ένας κανονισμός μη ευέλικτος που προτείνεται από την Κομισιόν και όχι οδηγία, αναγκάζοντας ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσουν μέρος του επιτυχημένου πλαισίου που έχουν και να το αντικαταστήσουν με κανονισμό, κανονισμό ευρωπαϊκό. Θα υπάρχει κόστος σοβαρό και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος. Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μείωση των προτύπων ασφαλείας εφόσον οι επαγγελματίες και επιθεωρητές ε, θα απομακρυνθούν από το βασικό τους έργο της εξασφάλιση της ασφάλειας. Το κόστος εφαρμογής της ε, νέας ε, πρόταση θα είναι περίπου 146 εκατομμύρια λίρες. Πολύ καλά. Έχουμε τις λίρες εδώ. Τις λίρες της Αγγλίας αυτή η πρόταση θα μπορούσε... Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω τι είχατε προηγουμένω. Αυτέ οι προτάσει θα μπορούσαν να μα οδηγήσουν ε, σε, ένα, ε, σε μια πολύ κακή κατάσταση νομική, καταστροφική. Ως Ευρωβουλευτής θα ήθελα να προτείνω το μοντέλο μας ασφαλείας στους συναδέλφους και θα ήθελα να βοηθήσουμε τις γνώσεις και την πραγματογνωμοσύνη μας για να ξανασυντάξουμε την πρόταση για να μπορέσουν να ωφεληθούν όλες οι χώρες. Ξέρω ότι πολλοί βουλευτές εδώ θα θελήσουν να επωφεληθούν από την πρόταση για να ζητήσουν μια διακοπή, μια αναστολή όλων των εξορίξεων σε ανοιχτή θάλασσα. Ζει όμως σε πραγματικό κόσμο και μέχρι το πράσινο λόμπι να μας παρουσιάσει μια βιώσιμη εναλλακτική στο πετρέλαιο και στο αέριο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μπορούμε να εξορίξουμε καλύτερα τους πόρους μας. Θα υποβάλουμε από την ομάδα μας πάρα πολλές τροπολογίες στο κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, για αυτήν την ε, ιδιαίτερα δροσιστική συμβολή από το Ηνωμένο Βασίλειο ο συνάδελφος Βίλτς που είναι παρόν ένας από τους δύο σκιώδεις συγητές που είναι παρόν η κυρία Βίλτς, συγγνώμη ευχαριστώ δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο ως Επιτροπή Περιβάλλοντος να υποβάλουμε μόνο γνωμοδότηση για την Ήτρε η Επιτροπή έκανε μια πρόταση για την ασφάλεια δραστηριοτήτων ανοιχτής θαλάσσης Πρώτα απ' όλα είναι θέμα ασφάλεια, ασφάλειας σε σχέση με τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές βλάβες και για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν και για τους ανθρώπους και για, για το ζωικό βασίλειο. Εμείς είμαστε η Επιτροπή. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε γιατί έχει να κάνει με την εξυγίανση των καταστάσεων και για το κλίμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με την Ήτρε. Δεν θα πρέπει μόνο εκεί να είναι αρμόδια. Φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο ευθύ εξ αρχή καθορίζεται η κατεύθυνση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ωστόσο, εκπεφρασμένα χαιρετίζω το ότι η Κομισιόν όσον αφορά την ε, δραστηριότητα στον τομέα αυτό προτείνει κανονισμό. Έτσι δίνεται στην Ένωση η δυνατότητα να επιβάλλει ελάχιστες προδιαγραφές στα κράτη-μέλη απευθείας. Φιλόδοξες προδιαγραφές σε επίπεδο ένωσης είναι περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε κοίτασμα είναι χρήσιμο για την απληστία των διαφόρων εταιριών. Προσπαθούν λοιπόν να αποκομίσουν κέρδη από κάθε τέτοια πηγή ανεξαρτήτως των κινδύνων. Και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει και η ζήτηση και οι τιμές. Πέρα λοιπόν από τις άμμους, πέρα από τα σχιστολιθικά, σχιστολιθικά προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε κοίτασμα και στο βυθό των θαλασσών, ακόμη και αν είναι χιλιόμετρα από την επιφάνεια των θαλασσών. Και η ίδια Κομισιόν γράφει στην πρότασή της ότι ο κίνδυνος ενός σοβαρού ατυχήματος από εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοιχτή θάλασσα είναι σοβαρός. Διαπιστώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι όντως η κίνδυνη αυτή δεν είναι θεωρητική. Εάν προκύψει λοιπόν ατύχημα, Πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι η υπεύθυνη εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει για όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να έχει δυνατότητα να το κάνει. Γι' αυτό το άρθρο 4 της πρότασης της Κομισιόν δεν μου φαίνεται αρκετά σαφές. Πρέπει σαφώς να καθοριστεί ότι υπάρχουν οι αναγκαίε οικονομικέ δυνατότητε για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι επιπτώσει πριν δώσουμε άδεια σε μια εταιρεία. Δεν θα πρέπει μόνο να παίρνουν τα κέρδη, θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρώσουν και για τις ζημίες. Προεδοποιώ, πρέπει να υπάρξει σημαντική αλλαγή τα αλλιώς θα πληρώσει ο φορολογούμενος. Πιστεύω λοιπόν ότι ο εισηγητής με τις προτάσεις του πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εξόριξη στην Αρκτική για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο δεν είναι σκόπιμη γιατί είναι πολύ ευαίσθητες αυτές τις περιοχές. Είτε η Αρκτική είτε ε, παρόμοιες περιοχές τόσο ευαίσθητες. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει για σοβαρό ατύχημα σε αυτές τις περιοχές. Καμία περιοχή σε τέτοιου τύπου περιβάλλοντα. Καμία συγγνώμη εταιρεία. Επίσης, ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ατυχήματα, αυτές οι εγκαταστάσει μολύνουν το περιβάλλον σε μικρές ποσότητες αλλά συνεχώς απορρίπτονται χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα Άρα αυξάνεται συνεχώ η μόλυνση. Ο, εάν δεν είναι σε θέση να σταματήσουν οι εταιρείε αυτή τη μόλυνση, δεν θα πρέπει να του χορηγούνται νέε άδειε, ιδίω σε ευαίσθητε περιοχέ. Οι εταιρείε αυτέ ένα μεγάλο τμήμα των επενδύσεών τους το κάνουν για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν νέα κοιτάσματα. Κλείνουμε τα μάτια στο ότι αυτές οι πηγές δεν είναι ανανεώσιμες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε αυτές οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας να στραφούν προς ανανεώσιμες πηγές παρά να προσπαθούν να εξορίξουν αυτά τα ορυκτά καύσιμα με όλο και υψηλότερο κόστος. Και ιδίω σε ευαίσθητες περιοχές πρέπει οπωσδήποτε να μην επιτρέπονται αυτές οι εξορίξεις και πρέπει να έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Θίξατε το θέμα γιατί δεν συμμετέχουμε ως Επιτροπή. Μπορώ να πω ότι πάλεψα για την Επιτροπή μας μέχρι τελευταίας ρανίδος. Αλλά τελικά στη διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε, των Επιτροπών αποφασίστηκε ναι, με δεν συμμερίζουμε πλήρω την άποψή σα, αλλά ε, βεβαίω τη συμμερίζουμε όσον αφορά τι αρμοδιότητε τη ε, Επιτροπή μα. Έχουμε βεβαίω ε, γνωμοδότηση να κάνουμε. Έχουμε ε, αποκλειστική αρμοδιότητα για κάποια άρθρα και από κοινού αρμοδιότητα για κάποια άλλα άρθρα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς ε, διαμάχης με τους συναδέλφους από την Ήτρε. Και εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή εδώ θα έπρεπε εμείς να είμαστε αρμόδιοι και όχι η Ήτρε, αλλά τέλος πάντων ε, πάρθηκε άλλη απόφαση. Το λέω εγώ ίδιο Νάλφο Ιβκο Χωρίς περιορισμό χρόνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέρυσι δεν ήμουνα στο Ευρωκοινοβούλιο, ήμουνα στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Και με τον τωρινό Πρωθυπουργό, τον Ζωα Μαρκερό, ήμασταν αντιπολίτευση. Αλλά είχαμε καταθέσει ένα νομοσχέδιο, έχω εδώ ένα αντίγραφο, για να απαγορεύσουμε την εκμετάλλευση ε, την υπεράκτη εκμετάλλευση σε μεγάλα βάθη. Λέγαμε ότι αυτό του είδους η εξόριξη υδρογονανθράκων είναι ε, ιδιαίτερα ενεργοβόρα, είναι ιδιαίτερα προβληματική. Πολλές φορές η οριζόντια Η οριζόντια γεώτρηση γίνεται σε πολύ μεγάλο βάθος και έχουμε και το πρόβλημα της Γουιάννα στα νυχτά της ε, Καγέν. Η Σέλη, το Τάλ και η Τούλο προσπαθούν ε, να ξεκινήσουν την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Η ΤΟΥΛΟ από μόνη της έχει μία πλατφόρμα ένσκο η οποία στοιχίζει 300.000 ευρώ τη μέρα. Στην Γουιάννα υπάρχει μια τεράστια βιοπικιλότητα που ευχαριστεί ιδιαίτερα την συνάδελφο Μπελιέ και όλους και υπάρχει ένα πρόβλημα για τις θαλάσσιες χελώνες. Φαντάζομαι ότι οι θαλάσσιες ε, χελώνες αξίζουν πολύ περισσότερο από ότι όλες οι offshore σε μεγάλα βάθη εκμεταλλεύσεις και γεωτρήσεις και παρά τις ενδιαφέρουσες προτάσεις της Κομισιόν και του εισηγητή θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί με αυτές τις εκμεταλλεύσεις. Πόσο μάλλον που για να έχει κανείς ενέργεια μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, όπως είπε και ο συνάδελφος Μπάς. Ευχαριστώ κύριε Κωσέ. Δεν σας είχα περιορίσει το χρόνο σας, όπως είπα. Έληξε η συζήτηση. να ζητήσω από την Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο και ευχαριστώ όσους υποστήριξαν την πρόταση της Κομισιόν και νομίζω ότι στόχος της Κομισιόν είναι σαφώς να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των πόρων αυτών που είτε το θέλετε είτε όχι θα παραμείνουν για πολλές δεκαετίες. Ακόμα και στον χάρτη πορείας 2050 για την ενέργεια, όπου εξετάζουμε σαφώς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, οι καλύτερες πηγές ενέργειας είναι βεβαίως οι ανανεώσιμες, αλλά πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές και ότι το πετρέλαιο και το αέριο θα είναι μαζί μας για πολλές δεκαετίες ακόμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να νομοθετούμε καταλήλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης επειδή υπάρχουν ορισμένες εξορίξεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι ορισμένες χώρες είναι πιο προχωρημένες από άλλες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η BP είναι πλάκη μια βρετανική ε, εταιρεία και είναι πράγματι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει σαφώς να ρυθμίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό έχουμε προτείνει έναν κανονισμό διότι θέλουμε να απευθυνθούμε απευθεία στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δραστηριοτήτων που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των δραστηριοτήτων. Είναι σαφές ότι η συζήτηση σχετικά με οδηγία ή κανονισμό θα λάβει χώρα σε αυτό το κοινοβούλιο και όπως ξέρετε η, Ήτρα, Επιτροπή Ήτρε προτείνει μια οδηγία και σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι εσείς υποστηρίζετε έναν κανονισμό και βεβαίως το Συμβούλιο φαντάζεστε ότι θα λάβει χώρα και λαμβάνει χώρα αυτή η συζήτηση περί της επιλογής σας. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και την υποστήριξη των βασικών γραμμών της πρότασής μας. Έχετε τονίσει ορισμένα θέματα τα οποία ε, πιθανόν ε, είναι δύσκολα και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τονίσατε τη σημασία τους, όπως επίσης ε, την χρηματική, την οικονομική υπευθυνότητα. Σήμερα οι ασφαλιστές δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις ζημιές που θα μπορούσαν να προέλθουν από τέτοια συμβάντα και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει και για το λόγο αυτό εξετάζουμε άλλες ε, πιθανές εναλλακτικές λύσεις και που βρίσκονται στην πρότασή μας. Κατανοούμε ε, την ανησυχία σας. Ε, Βεβαίω ξέρετε ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις σε αυτό το στάδιο. Υπήρξε επίσης μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έκανε ο εισηγητής, δηλαδή η δηλαδή κοινή επιθεώρηση από κράτη-μέλη σε δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλος. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα την εκτιμήσει αυτή την πρόταση αλλά είναι αληθές και έχουμε άλλα παραδείγματα όπου σαφώς υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες ε, που δεν αφορούν μόνο ένα κράτος μέλος ε, και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερη περιφερειακή συνεργασία στον τομέα αυτό. Θα ήταν χρήσιμο αυτό. Έχουμε επίσης όπως καταλάβατε ε, το θέμα της ε, διάλυσης, της αποσυναρμολόγησης των πλατφορμών και των εγκαταστάσεων που είναι ένα σημαντικό θέμα που κανονικά θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην συμφωνία διοδότησης και στην άδεια, στην παραχώρηση στον φορέα εκμετάλλευσης. Να υπάρξει δηλαδή όλος, να περιλαμβάνεται όλος ο κύκλος, όλη η διάρκεια ζωής και η διάλυση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο τονίσατε, είναι ο ρόλος της ΕΜΣΑ, της Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Ο κανονισμός για την ΕΜΣΑ πρόσφατα διευρύνθηκε, επεκτάθηκε για να επιτρέψει στην ε, υπηρεσία ΕΜΣΑ να εμπλέκεται ε, σε υπηρεσίες εξόριξης ανοιχτής θάλασσας και βεβαίως αυτό δεν προχωράει τόσο πολύ όσο πολλοί από εσά θα ήθελαν, δηλαδή η εποπτεία από την ΕΜΣΑ. Δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος της ΕΜΣΑ, δεν είναι ακόμη ο ρόλος της ΕΜΣΑ και ίσως ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί βήμα προς βήμα προοδευτικά. Η Κομισιόν δεν πάει τόσο μακριά ως προς τη διαφάνεια. Βεβαίως αυτό αποτελεί μέρος της πρότασής μας και χαιρετίζουμε ε, ιδέες για την βελτίωση της διαφάνειας σχετικά ε, με τα ευαίσθητα θέματα θα πρέπει να το δούμε επίσης στη διαδικασία αδειοδότηση. Ήμουν στην Νορβηγία πριν ε, λίγο καιρό. Ενδιαφέρεται από την Αρκτική η Νορβηγία και η Νορβηγία είναι χώρα η οποία εξετάζει εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό και έχουμε εμπιστοσύνη διότι η Νορβηγία θα θέσει τους απαιτούμενους όρους για να ε, ανοίξουν νέες οδοί στην Αρκτική για εξόριξη. Νομίζω ότι τεχνικά είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να ρυθμιστεί στο επίπεδο της αδειοδότησης που θα είναι και καλύτερο προληπτικό μέτρο σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες, διότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο θέμα. Θα σταματήσω εδώ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολλές τροπολογίες σε αυτή την Επιτροπή. Η Επιτροπή Ήτρε θα συζητήσει το θέμα αυτό αύριο το πρωί και είμαι βέβαιος ότι οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο θα είναι ενδιαφέρουσες. Προσβλέπουμε σε αυτές με μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζουμε να έχουμε και πρόοδο στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Εργαζόμαστε εδώ και 6 μήνες για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και περιμένουμε εφόσον πρόκειται για προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας να μπορέσουμε να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πριν το τέλος του έτους, διότι αυτό είναι το θέμα εδώ, είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την εξερεύνηση και παραγωγή στην ανοιχτή θάλασσα και έχουμε έναν κοινό στόχο την δημιουργία των καταλήλων συνθήκων και ε, νομίζω ότι σε αυτό αποβλέπει και το σχέδιο. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Οπότε κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. 12 Ιουλίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 6 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου. Α, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα της διάταξης. 17 και 18. Θα τα συζητήσουμε μαζί. Πρόγραμμα έρευνας καινοτομίας ορίζοντα 2020 και το ειδικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του ορίζοντα 2020. να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κρίστιαν Σίλβιου Μπουσόη. Σωστά το πρόφερα. Μπουσόη. Πολύ καλό, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους σκιώδεις και τα μέλη για τις τροπολογίες, περίπου 400 για τον κανονισμό και 200 για τις εφαρμοστικές αποφάσεις του 2020, ορίζω 2020. Θα αναφερθώ σε μερικές σημαντικές τροπολογίες. Ίσως όχι όλες, αλλά δεν είναι ίσως η τελική μου τοποθέτηση, γιατί οι επιπτώσεις κάποιων τροπολογιών χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Και θέλω να ακούσω και τους συναδέλφους μου, που θα υποστηρίξουν τις τροπολογίες τους. Πολλές τροπολογίες εισάγουν νέε ιδέες, όπου το, αθνικό, το αρχικό μου σχέδιο δεν τροποποιούσε την πρόταση της Επιτροπής. Με χαρά θα τις υποστηρίξω. Κάποιες τροπολογίες θεωρούν, ε, ασχολούνται με την ελκυστικότητα του προγράμματος για τους ερευνητές. Πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπα και σε προηγούμενη συζήτηση, είμαι υπέρ ε, μιας οριζόντιας προσέγγισης, δηλαδή να εμπλέκονται διάφοροι τομείς της επιστήμης. Είναι βασικό αυτό. Για τα βλαστοκύτταρα πολύ λεπτό θέμα. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Είναι τομέα όπου θα επιχειρήσω να προτείνω κάποιους συμβασμούς ή έναν. Μερικές τροπολογίες είναι πιο φιλόδοξες από την πρόταση Επιτροπής, άλλες είναι πιο περιοριστικές. Και εγώ υπέβαλα τροπολογίες που ε, κάπως αλλάζουν ε, την διατύπωση για να λάβω υπόψη τις προτάσεις επιτροπής. Όταν μιλάμε για εναλλακτικέ στα ε, εμβρυικά βλαστοκύτταρα δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεκριμένοι να αφήνουμε δυνατότητα και για νέες ε, προσεγγίσεις. Να μην περιζόμαστε μόνο στο αίμα από τον πλακούντα και τον ομφάλιο λόρο. Θα ήθελα να πω ότι αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μάλλον να δώσουμε ένα συγκεκριμένο να τυποποιήσουμε αυτά τα κύτταρα του, ε, των εμβρίων. Τότε μπορούμε να εξετάσουμε άλλε εναλλακτικέ λύσει. Μιλάμε επίση, πολλέ τροπολογίε μιλάνε για τι νανοτεχνολογίε. Πολύ σημαντικό. Φυσικά οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και τι επιπτώσει στο περιβάλλον. Όμω αυτό το θέμα, η πτώση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία είναι μια πρόκληση. Μου αρέσουν μερικές τροπολογίες της ε, κυρίας Γκουτιέρεθ Κορτίνα στις, ε, για τις βιοτεχνολογίες, ιδίως για τις επιπτώσεις στη γεωργία, για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Βεβαίως, θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματική χρήση των ε, ενεργειακών πόρων, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται χωριστή προτεραιότητα για την οικοκαινοτομία. Η οικολογική καινοτομία είναι πολύ ευρία έννοια περιλαμβάνει πολλέ δραστηριότητες που ήδη καλύπτονται σε άλλους τομεί. Το τμήμα της υγείας. Μας ενδιαφέρουν οι χρόνιες ασθένειε. και η πρόληψη και άλλα θέματα συμπληρωματικά σε αυτά που έχω ήδη προτείνει και φυσικά θα τα υποστηρίξω. Ενδιαφέρουσες επίσης τροπολογίες υπάρχουν για την έρευνα στην ε, ε, σχέση φίλου με την ε, ε, εκδήλωση κάποιων ασθενειών. Κάποιες τροπολογίες όμως δεν με βρίσκουν τόσο σύμφωνο. Είναι αυτές που μιλάνε πιο συγκεκριμένα για μια κατηγορία ασθενών ή κάποιες που προσθέτουν και άλλες ασθένειες, τις χρόνες ασθένειες που πρέπει να χρηματοδοτούνται. Ο συνάδελφος μου Λουχάν από τη Ρουμανία αναφέρεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες στον τομέα της ε, υγείας δεν νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα. Θα προτιμούσα το κείμενο να είναι γενικό. Αυτό ανοίγει την, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και για δραστηριότητες που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τις χρονικές, χρόνιες ασθένειες. Καλύτερα θα ήταν να διαγράψουμε όλα τα παραδείγματα. Όλες οι χρόνιες ασθένειες να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Καμία να μην θεωρείται ότι εξαιρείται. Μερικές τροπολογίες ε, προσθέτουν παραδείγματα. Θέλω να το αποφύγω. Αλλά ελπίζω να ε, υπάρξει συμβαστική λύση. Με ενδιαφέρουν και συμφωνώ οι περισσότερες άλλες τροπολογίες για τις σπάνιες ασθένειες. Σημαντική προτεραιότητα. Επίσης, θέματα, τα θέματα της γονιμότητας, ε, της παρέμβασης στην συμπεριφορά των ανθρώπων και άλλα θέματα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στη διατύπωση για τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Για την επιστηστική ασφάλεια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που έβαλαν τροπολογίες για την αλυσίδα προσφοράς και τις επιπτώσεις του περιβάλλον. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις αλυσίδες ε, προμήθειας και να προωθήσουμε καλύτερη διατροφή για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας για την ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε, τι στόχους θα θέσουμε για να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, αν και δεν είναι εδώ το κατάλληλο κείμενο για ιδεολογικές συζητήσεις, αλλά είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας. Άρα σημαντικό και να το συζητήσουμε. Ο Horizon 2020 πρέπει να συμβάλλει και στην αύξηση χρήσης ανανεώσιμων, αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας, και επίσης λύσεις αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες. Γι' αυτό πρέπει να συμβάλλουμε στους περιβαλλοντικούς μας στόχους μέσω αυτού του προγράμματος Horizon 2020. Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν δράσεις για τα ύδατα, διαχείριση υδάτων, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και τα περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα. Αλλά να δούμε ποιος θα είναι ο ακριβής τίτλος. Συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι προκλήσει των κοινωνιών πρέπει να συζητηθεί περισσότερο. Υπάρχουν διάφορα ποσοστά που προτείνονται, υπάρχουν ερωτήματα και επί της αρχής για το γιατί θα πρέπει ορισμένα χρήματα να πηγαίνουν ειδικά και αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μιλήσω τώρα γενικά για τον προπολογισμό. Πρότεινα μια τροπολογία όλα τα ποσά να γίνουν ποσοστά. Το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μου αυτό μας εγγυάται ότι ό,τι διαπραγματεύσει και να γίνουν για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα διατηρηθεί το σχετικό βάρο εντό του προγράμματος κάθε τομέα. Είναι σημαντικό αυτό. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσετε σε αυτή την αρχή. Το συζητήσαμε στην Ήτρε και συμφωνήσαμε που είναι η επί της ουσίας αρμόδια. Επί των στοιχείων έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά ελπίζω να καταλήξω συμφωνία. Θα υποστήριζα αύξηση του συνολικού προϋποτολογισμού και θα ήθελα να αυξηθεί η έρευνα για την υγεία, προϋπόθεση για ανταγωνιστικότητα και ευημερία μακροπρόθεσμα. Επίσης, για τον προϋπολογισμό Θα ήθελα ο προπολογισμό να είναι συνολικά πιο ισορροπημένος. Για το εάν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας να διαχειρίζεται αποκλειστικά τον προπολογισμό, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποια χρήματα να μπουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την βιομηχανική πρωτοπορία. Βεβαίω και η θεμελιώδη έρευνα είναι βασική, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για ενέργειε που να έχουν ω επίπτωση καινοτόμα προϊόντα. Όχι υπερβολική χρηματοδότηση τη θεμελιώδου έρευνα που δεν καταλήγει πάντα σε καινοτομία. Μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ θα λάβετε την πρότασή μου για να είναι σαφώ κείμενο στο τέλο στη διάθεσή μα. να κάνουμε όσο χρειάζεται συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών για να συζητήσουμε τους συμβασμούς. Όμως, ευθύς εξ αρχής, να τονίσω ότι το κείμενό μου θέλω να είναι αρκετά σύντομο, να μην είναι ένα συνονθήλευμα όλων των στοιχείων που θα έχει αναφέρει ο καθένα. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, κύριε Μπουσόη, για την αναλυτική παρουσίαση της έκθεσής σας οι σκιώδεις ηγητές. ΕΛΚ. Η κυρία Κουτιέρεθ Κορτίνε. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη για την προσπάθειά του και να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι τα προηγούμενα. Εμείς έχουμε εργαστεί για το πέμπτο, για το έκτο πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και πρέπει να σας πω, δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να καταφέρει να διαβάσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό, η ανάγνωση αυτού του προγράμματος ισοδυναμεί με, με, με μια πάρα πολύ δύσκολη εξέταση ενός πανεπιστημιακού μαθήματος. Και πολλές φορές με ανησυχεί εδώ αυτό το τεχνικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει. Δηλαδή, έχουμε εμεί μια γενική περίληψη του προγράμματος και μετά πάνω σε αυτήν τη γενική περίληψη κατατίθενται τροπολογίες. Οπότε πραγματικά προσοχή με τις συμβαστικές τροπολογίες διότι στο κάθε κεφάλαιο ανταποκρίνεται κάτι το πολύ συγκεκριμένο, στο κάθε κεφάλαιο έχουμε έναν οργανισμό που το διαχειρίζεται. Οπότε πρέπει να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχεία. Καλύτερα να επαναλαμβάνει κανείς τέσσερις φορές το ίδιο πράγμα και να ψηφίζει τέσσερις τροπολογίες παραπάνω, από ότι να έχουμε την παράληψη. Το Συμβούλιο αποφάσισε όλη αυτή την ιστορία μετά από πιέσεις ιταλικές που εγώ δεν θέλω τώρα να σας αναφέρω, δεν θέλω να ξεκινήσω τέτοια ιστορία. Αλλά τα πράγματα δεν μπορούν να μετατοπίζονται μέσα στην έκθεση γιατί άπαξ και αλλάξουμε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο πρόγραμμα πάνε τα πάνω κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γενικό να περνάει μέσα από το ειδικό. Εμείς έχουμε ζητήματα που αφορούν στον ορίζοντα, ορίζοντα, στον ορίζοντα 2020. Ας πούμε ο ορισμός του τι εστί υποδομή. Μιλάμε δε για υποδομές και όλοι κατευθείαν τρέχουν στα διαρθρωτικά ταμεία. Όχι, οι υποδομές δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως. Υπάρχουν και υποδομές που είναι εντελώς διαφορετικού τύπου για την κλιματική αλλαγή, για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Στον ορίζοντα 2020 η ίδια αντίληψη έχει διαφορετικούς ορισμούς στο λεξικό. Χρειάζεται κανείς να γνωρίζει ε, τις εξισώσεις για να μπορεί να το καταλάβει. Και ξέρετε τις εξισώσεις πια δεν τις διδάσκουμε, δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ξεπερασμένες. Πρέπει λοιπόν εμείς να ανησυχούμε ιδιαίτερα για όλη αυτή τη γενική αντίληψη. Για το περιβάλλον θέλω να επιμείνω σε δύο-τρία πράγματα. Η πόλη είναι ένα αστικό τοπίο. Κατά συνέπεια είναι περιβάλλον. Και όταν εμείς μιλάμε για, πισικούς, για, μιλάμε για πολιτιστικούς πόρους, αυτό ισχύει και για, τις, την πόλη ή για ένα παλιό ρηχείο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε, να βάλουμε πάρα πολλά στοιχεία, γιατί την αηφορία πρέπει να την προστατεύσουμε συνολικά για το σύστημα του νερού εγώ βέβαια δεν έχω πλήρη εικόνα της κατάστασης, αλλά διαπραγματεύομαι και συζητώ συχνά με τεχνικούς ή με επιχειρήσεις σχετικά. Η τεχνολογία για το φιλτράρισμα των νερών έχει προχωρήσει πολύ, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα για το τι εστί ο ιδρικός κύκλος, δηλαδή τι γίνεται με τη βροχή κτλ. Πρόκειται λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον κύκλο του ύδατος. Όπως επίσης πρέπει να ελέγξουμε και τις πηγές και τα φρεάτια. Διότι ξέρετε ότι η λεκάνη και τα, και τα φρεάτια είναι πολύ ευρύτερα από ότι η λεκάνη του ποταμού του Ιδίου. Υπάρχει μία μελέτη για τις πηγές ε, και για τα υπόγεια ύδατα του, ε, του, ε, του Δούναβη που επηρεάζουν τις περισσότερες χώρες από, ότι, από αυτές που διατρέχει ο ποταμός. Δηλαδή αν αρχίσουμε εμείς και πειράζουμε τις όχθες του Δούναβη, επηρεάζουμε τους ιδρικούς πόρους και άλλων χωρών. Όλες οι τεχνολογίες χρειάζονται όχι μόνο για τις νότιες χώρες, αλλά χρειάζονται για να μπορέσουμε, για να, μπορέσουμε να διορθώσουμε ε, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις ζημιές. Υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά ζημιώνουν το περιβάλλον και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και τώρα για την μελλοντική γεωργία δεν έχουμε κάνει ακόμη την αγροτική μας επανάσταση που απαιτεί κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται έρευνα για νέα φυτά που είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα. Ε, δεν μπορούμε εμείς ακόμη να, φυτεύουμε μαρούλια στο νότο που, παίρνουν, που πίνουν ένα σωρό νερό ενώ θα μπορούσαμε να φυτεύουμε κακτοειδή. Αλλά αυτά τα κακτοειδή βρίσκονται στα εργαστήρια των πανεπιστημίων. Μόνο το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε αυτή την έρευνα. Η νέα ατζέντα λοιπόν της γεωργίας θα πρέπει να είναι ένα χρονοδιάγραμμα που θα εισακούει τις κλιματικές αλλαγές. Και τώρα κοιτάστε, σας το λέω έτσι και καλαμπορίζοντας. Είναι σαν τον καθηγητή που θεωρεί ότι το δικό του το μάθημα είναι και το πιο σημαντικό. Αλλά δείτε τι γίνεται για την ε, διαφάνεια. Το σύστημα πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και δυσνόητο και θολό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο κώδικας για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα και το public assert και το public data θα πρέπει να δούνε τι γίνεται με τις δημοσιεύσεις. Σήμερα οι ερευνητές για να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό πρέπει να πληρώνουν τη δημοσίευση και μετά πρέπει να ξαναπληρώνουν για να αγοράσουν το περιοδικό με τις δικές τους δημοσιεύσεις. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν, ε, δεν έχουν εισοδήματα για να αγοράζουν ε, κονδύλια για να αγοράζουν πίσω αυτά τα περιοδικά για τις ε, βιβλιοθήκες τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά θα πρέπει να λυθούν. Όποιος δημοσιεύει, ας δημοσιεύει τα στοιχεία τώρα της έρευνας πρέπει πολλές φορές να κρατούνται μυστικά όπως και η καινοτομία. Δεν θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις έναν ερευνητή για να δημοσιεύει μετά αυτό το οποίο ερεύνησε για την επιχείρηση. Πρέπει να υπάρχει το public access access και, το public, το, τα, και τα public data. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ μυστικού και δημοσίου. Και δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός όπου τελικά εσύ πρέπει να πληρώνεις για να αγοράσεις τη δική σου δημοσίευση. Και τα public data επίσης για βασικές έρευνες άνοιχτες ή για καινοτομία. Ο Βιτόριο Πρόντι. Πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Α, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για όλη αυτή την τεκμηρίωση που είναι πολύ σημαντική και δεσμευτική. Πιστεύω όμως ότι τα δύο θέματα είναι πολύ παρεμφερή. Οπότε ή θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε σαφώς ή να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο έγγραφο, διότι εδώ έχουμε ιδέες, αντιλήψεις που επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές. Και οι τροπολογίες κατατέθηκαν και στα δύο έγγραφα και πολλές φορές κουραζόμα... Ε, δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε και να αξιοποιήσουμε πλήρως το καθένα από τα δύο έγγραφα. Ας πούμε το establishment και η implementation του εγγράφου του ιδίου. Εμείς έχουμε εγγραφά τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ σημαντικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ παίζεται η δική μας ικανότητα ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να πετύχουμε να βρούμε την αριστεία. Και για τα θέματα που αφορούν στην Επιτροπή μας Έχουμε να ασχοληθούμε με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Για τη δημόσια υγεία Έχουμε τεράστιες δυνατότητες και πρέπει να τις αναγνωρίσουμε. Και αυτές οι δυνατότητες τονίζονται στις ε, τροπολογίες, αλλά τα γενώματα και τα τοξώματα είναι απολύτως απαραίτητα για αυτήν την ειδική ιατρική που περνάει μέσα από την πλήρη αναγνώριση του γονοδιώματος του ε, ασθενή για να μπορέσει να πετύχει να, να, να πετύχουν ιδιαίτερες θεραπείες στον ασθενή. Διάβαζα χθε το International Herald Tribune για τη θεραπεία μιας οξείας προχωρημένης λευκαιμίας που στάθηκε δυνατό να θεραπευθεί, διότι ο ότι για τον ασθενή αυτό κινητοποιήθηκε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο της πολιτείας της Ουάσιγκτον που έκανε αυτήν την χαρτογράφηση του γονοδιώματος με πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και είναι εξίσου σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Τώρα, κάτι που πάει παράπλευρα. Για τη χορήγηση αδειών για τη χρήση αυτών των φαρμάκων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τον πειραματισμό μεθόδους που να μην χρειάζονται πειραματόζωα, αλλά να μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, κυταρική καλλιέργεια. και να μπορέσουμε να αποφύγουμε και τον κίνδυνο της αναποτελεσματικότητας του φαρμάκου. Πολλές φορές οι εταιρείε πίσω από όλη αυτήν την ιστορία των πειραμάτων των φαρμάκων, χαρακώνονται πίσω από την ιστορία πειραμάτων στα φάρμακα για να δικαιολογήσουν την υψηλή του τιμή. Εμείς ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις τεχνολογίες που χρειάζονται για τη χορήγηση αδειών για τα φάρμακα, έχοντας ως κριτήριο και τη μείωση του κόστους και την μεγαλύτερη ακρίβεια των δοκιμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως εξίσου σημαντικό, σημαντική είναι και η πορεία ε, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ετέθη το πρόβλημα του νερού. Φυσικά το νερό είναι πολύ σημαντικό, αλλά εμείς μπορούμε και πρέπει να επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο σκεπτικό για όλους τους φυσικούς πόρους. διότι εν δυνάμει έχουμε πολλούς άλλους φυσικούς πόρους που μπορούν να εκλείψουν περισσότερο από ότι το νερό. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε μαζί με τον εισηγητή και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, Βιτόριο. Επόμενος. Επόμενη, η Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητής έκανε σημαντική εργασία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό και όλοι αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ιουαλία έχουμε 84 ε, εκατομμύρια για έρευνα, χρηματοδότηση για έρευνα ε, που δεν ωφελούν ε, μόνο την υγεία αλλά προσφέρουν ε, δυνατότητες σημαντικές αναπτυξιακές και θα ήθελα το πρόγραμμα Horizon 2020 να βασιστεί στην εργασία που έγινε στο παρελθόν να να συμβάλλει σε αηφόρο οικονομία. Όπως ανέφεραν ορισμένοι προλαλήσαντες, είναι επίσης το θέμα υγείας είναι σημαντικό, αλλά θα ήθελα να εσταθώ στο τελευταίο σημείο που ανέφερε ο κύριος Πρόντι για την κλιματική κλιματική Αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, νομίζω ότι για αυτήν είναι κρίσιμο να εξετάσουμε πώς το χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση της κλιματικής αλλαγής, την μείωση της ρήπανσης, την διατροφική ασφάλεια, την υγεία. Ε, είναι σημαντικά τα θέματα αυτά, όπως και η υγεία. Η έρευνα είναι αναγκαία ε, για την ε, διατροφική αλυσίδα ε, και για τα προϊόντα που παράγονται και τα συναφή θέματα θα πρέπει ε, το σχέδιο γνωμαδότησης ε, να αναφερθεί περισσότερο σε αυτούς τους στόχους. Αναφέρθηκε ο εισηγητής σε διάφορα θέματα, αλλά ε, εστιαστήκαμε στο να ενισχύσουμε ορισμένα άλλα θέματα. Ίσως η αηφορία είναι σημαντική και πρέπει να εξετάσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο της χρηματοδότησης επίσης. Ένα μια από τις προτάσεις που κάναμε στην Επιτροπή είναι να κάνει ε, μια μελέτη, ε, μια αξιολόγηση κοινωνική και οικονομική και αηφορίας ε, για ορισμένα έργα. Δεν πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα όπως το ITER ή την ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, ένα σύστημα, καλύτερα ένα σύστημα πληροφορίας παρακολούθησης που σημαίνει περισσότερη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς που εργάζονται στον τομέα σε διεθνή βάση και είναι ουσιαστικό οι προτεραιότητες οι ερευνητικές να αποφασιστούν σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών επίσης. Γι' αυτό προτείναμε τροπολογίες που προτείνουν διάλογο, πλατφόρμες διαλόγου για το σκοπό αυτό. Ε, Παραδείγματο χάρη για μικρούς ε, αγρότες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην καινοτομία. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να αναγνωριστεί κυρίως στα πλαίσια της διατροφικής αλυσίδας και για να χρησιμοποιηθούν τοπική παραγωγή κυρίως σε σχέση με την καλή διαβίωση των ζώων. Το άλλο σημείο είναι η ευθυγράμμιση σχέσης ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία. Η συνδυασμός αυτών των ταμείων αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της έρευνας και της καινοτομίας. Πιστεύω ότι μπορούμε ε, από αυτήν την Επιτροπή να κάνουμε μια δήλωση ισχυρή για το ορίζον 2020 για να συμβάλλουμε ε, σε αηφόρο ανάπτυξη και σε μια ε, οικονομία όπου θα γίνεται αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές. Σούσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σε αυτή την έκθεση για την έρευνα και την καινοτομία ορίζοντας 2020 είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά παγκόσμια. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ικανότητά του για ένα θέμα τόσο δύσκολο και τόσο πλατή. Και, αυτό πέρα από τις ε, διαφορές απόψεων που μπορούμε να έχουμε με τον εισηγητή. Θέλω να σταθώ τώρα στις τροπολογίες που κατέθεσε η ομάδα μου, η Γκουέ, για το θέμα της υγείας. Έχουν κατατεθεί τροπολογίες από την κυρία Λιωτάρ, που είναι η, η, η συντονίστρια 343 και 346 που αφορούν στις ίσες ευκαιρίες και στις μεταφορές και έχουμε και τις τροπολογίες που έχω καταθέσει εγώ και που αφορούν σε διάφορα σημεία. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, λήψεις ε, στις ε, επενδύσεις για, τις, για την ερεύνα των ασθενειών. Επίσης υπάρχει ανικανότητα έρευνας σε, σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ε, πανδημίες. Επίσης, για την παροχή φροντίδας και θεραπείας στους πολίτες και στους φτωχούς. Πιστεύω ότι γι' αυτά μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που θέτουν προβληματικά. Κατέθεσα την τροπολογία αριθμός 53, η οποία αφορά στα βλαστοκύτταρα. Η Κομισιόν λέει ότι δεν χρειάζεται άδεια για τα βλαστοκύτταρα. Για τη δημιουργία δημοσίων ανοιχτών τραπεζών για τα βλαστοκύτταρα. Μετά κατέθεσα την τροπολογία 130 η οποία διαφωνεί με τον εισηγητή και θα πρέπει να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε. Για αυτό το σημείο προτείνω οι προτεραιότητες για την έρευνα και τη χρηματοδότηση να γίνονται βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων. Ορίζοντας 2020 λέμε εμείς δεν μπορούμε εμείς σήμερα στο 2012 να υποβάλουμε προτάσεις αγνοώντας ε, το ποιες θα είναι οι προτάσεις που θα προκύψουν από την πρόοδο μέχρι το 2020. Οπότε εμείς πρέπει να προβλέψουμε αυτήν την πρόοδο. πρόοδο. Προοδεύουμε ανάλογα με την εξέλιξη της γνώσης. Τώρα μια άλλη παρατήρηση. Η ομάδα μου είναι ανοιχτή για τη διαπραγμάτευση συμβιβαστικών τροπολογιών με τον εισηγητή. Θέλω όμως να αντιδράσω σε κάτι που άκουσα εδώ. Ο κύριος Πρόντι νομίζω το είπε. Μίλησε για εξατομικευμένη ιατρική. Εγώ έχω αμφιβολίες. Διότι δεν έχουμε επιστημονική απόδειξη για κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Δεν πρέπει εμείς να δημιουργούμε φρούδες, ελπίδες για την εξατομικευμένη ιατρική. Απέχουμε παρασάγκας από αυτό. Αν ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες πενεύουν ε, τα επιτεύγματά τους, είναι καθαρή προπαγάνδα. Πετσελίζα, ευχαριστώ τον Σάλφα Μπουζό για την εργασία και την ε, καλή διάθεση που έδειξε να συμπεριλάβει στις περαιτέρω συζητήσεις ε, τι απόψει που θα εκφραστούν. εκφραστούν. Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα ατελείωτο κατάλογος ασθενειών. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πού είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη ασκία, αξία. Ξέρω ότι στην Ήτρε, στις συζητήσεις για την υγεία, δίνεται προτεραιότητα στην ε, ευρωπαϊκή έρευνα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι εθνικό θέμα η έρευνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε για την έρευνα. Είναι προϋπόθεση γιατί οι ασθένειες είναι παγκόσμιες βέβαια. Ε, εντός κάποιων κρατών είναι πολύ λίγες περιπτώσεις και οι σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών, οι σοβαρές ασθένειες των παιδιών, ιδιαίτερα όταν είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας είναι δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρξουν ειδικέ διατάξεις για χρήση κάποιων ε, φαρμάκων και αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε και κάποια έρευνα και για τα δύο λοιπόν αυτά θέματα, σοβαρές ασθένειες και σοβαρές ασθένειες των παιδιών, πάντα η θέση του Κοινοβουλίου ήταν στο έκτο και το 7ο πρόγραμμα ε, πλαίσιο. Δεν τα επιβάλαμε βέβαια όσο θα θέλαμε, αλλά εδώ θα πρέπει να επανέλθουμε και παρακαλώ να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες μου για το θέμα αυτό και να τις υποστηρίξουμε. Επίσης υπέβαλα τροπολογίες που αφορούν το θέμα διάγνωση και θεραπεία. Αν διαβάσουμε τη γράφη επιτροπή, δημιουργείται η εντύπωση, δεν θεωρώ ότι γίνεται για λόγους κακών προθέσεων, αλλά θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι παράγονται μεγάλες ποσότητες στοιχείων Έχουμε δυνατότητες να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί κάποια ασθένεια, αλλά τι χρησιμεύει αυτό στον ασθενή. Να ξέρει ο ασθενή ότι θα είναι αυτέ ή όχι επιπτώσει είναι θέματα. Υπάρχουν ασθένειε όπου δεν υπάρχει θεραπεία, δεν έχουμε καμία δυνατότητα πρόληψη. Γι' αυτό το θέμα διάγνωση να συνδυαστεί με το θέμα πρόληψη και θεραπεία. Τι σχέση έχει τι όφελος έχουμε από, τον, από την διάγνωση, τη σωστή διάγνωση, εάν δεν μπορεί να μας βοηθήσει για την πρόληψη και τη θεραπεία. Πρέπει λοιπόν η προτεραιότητα να είναι σε αυτή τη σύνθεση. Δηλαδή η διαδικασία διάγνωσης να μας χρησιμεύει για να εξάγουμε θεραπευτικές επιπτώσεις, συμπεράσματα. Το είπε και ένας προηγούμενος συνάδελφος και υποστηρίζω και αυτό που είπε ο Βιτόριο Πρόντι για την εξατομικευμένη ιατρική. Πρέπει λοιπόν να το υποστηρίξουμε αυτό. Κάτι ιδιαίτερο. Πρόληψη. Για τους ανθρώπους. Για τους άνδρες μάλιστα. Όλα τα θέματα που αφορούν την πρόληψη της ε, παρενέργειας υπάρχουν πολλές παρενέργειες ε, πολύ βαριές Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που εργάζονται για την πρόληψη, για τους άνδρες και θεωρούν ότι χρειάζεται μία όθηση από την πολιτική. Τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά χρειάζεται περισσότερη όθηση από πλευράς πολιτικής. Θα μειώνονταν πολλά προβλήματα. Τελευταίο, για τα βλαστοκύτταρα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για το θέμα αυτό. Τις διάβασα πολύ προσεκτικά πολύ από το ΕΛ και στην Ήτρε υποστηρίζουν τη γραμμή Νικολάζου, Ξαμπόρσκα και άλλων. Υπάρχουν και νομικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Προσπάθησα με βάση αυτά που είπε ο Σάνθος Μπούζοη να καταλήξω σε κάποια συμβαστική πρόταση που από τη μία να υποστηρίζει την ιδέα του κ. Μπούζοη εναλλακτικέ δηλαδή ε, έρευνες να μην έχουμε μία ή δύο μόνο εναλλακτικέ, αλλά και τι άλλε εναλλακτικέ που θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε στο μέλλον να τι υποστηρίξουμε. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να εμπλακούμε στην ε, διαμάχη για το εάν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έρευνα ή όχι. Δεν θα υπάρξει συμβασμός με ευρεία υποστήριξη. Θα υπάρξουν πολλές διαμάχες, πολλή ανησυχία για το θέμα αυτό θα πρότεινα λοιπόν, επειδή έχουμε πάνω από 600 τροπολογίες, είπαμε πριν ξεκινήσει τη διαδικασία ότι θα ασχοληθούμε με τις βασικές μας αρμοδιότητες. Υγεία, περιβάλλον, προστασία των τροφίμων. Θα έπρεπε νομίζω να το βγάλουμε απ' έξω το θέμα αυτό. Να πούμε ότι οι τροπολογίες αυτές να συζητηθούν στην Ήτρε και στη Γιούρη που είναι αρμόδιες. Ότι δεν θα αναλωθούμε με τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν θα φθαρούμε. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να υπάρξει συμβασμό. Είναι μόνο γνωμοδότηση το δικό μα κείμενο. Δεν είναι βασική αρμοδιότητά μα. Αρμόδιες για τα ηθικά και τεχνικά θέματα είναι οι άλλε επιτροπές. Ίσως ήταν λοιπόν σκόπιμο να μην ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πέτερ Λίζε. Γιούντιτ Μέρκης. Ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους ε, για την ε, παρουσίαση όλων των θέσεων. Ορίζοντας 2020 είναι η τρίτη γραμμή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα τεράστιο κονδύλιο, ένα τεράστιο ποσό για την αναζωγόνηση της, νέας, της οικονομίας μας. Πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όμως αυτό το κονδύλι κατακαιρματισμένα, διασκορπίζοντάς το σε διάφορους στόχους, χωρίς να λέμε ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσουμε ή θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα, επικεντρούμενοι επί των στόχων επιτρέποντας την συγχρηματοδότηση είτε του ιδιωτικού τομέα είτε της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές το ψάχνουμε πολύ, διαχαιόμαστε χωρίς να είμαστε ακριβείς στο τελικό μας αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε τρεις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Δημογραφικό πρόβλημα, Έχουμε τη γύρανση του πληθυσμού με την ασωρό αρρώστιες που συνδέονται με αυτό. Έχουμε το πρόβλημα της κινητικότητας ε, και χρειαζόμαστε για όλα αυτά να βρεθούμε λύσεις όπως επίσης χρειαζόμαστε και μια δίκαιη οικονομία. Αν εμείς είμαστε ιδιαίτερα περιγραφικοί και λεπτομερείς όλα αυτά τα οποία λέμε ε, συνδέουμε όλα αυτά τα ζητήματα το ένα με το άλλο. Θα έπρεπε λοιπόν να ξεκόψουμε αυτόν τον δεσμό και να δώσουμε το κάθε θέμα μεμονωμένα. Τώρα για την έρευνα. Υπάρχει πρόβλημα στην έρευνα με υπηρεσίες και καινοτομία για τα αποτελέσματα της έρευνας. Χρειάζεται μία όθηση στην οικονομία μας. Χρειάζεται ανάπτυξη, απασχόληση. Εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη σπροξιά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να βγούμε μέσα από αυτό το θανατηφόρα διέξοδο. Χρειάζεται συγκεκριμένο, χρειάζεται όχι μόνο η γνώση αλλά η εφαρμογή αυτής της γνώσης. Επίσης, για την καινοτομία μπορούμε να τη, χρησιμοποιήσουμε ως κινητήρα. Δεν πρέπει όμως να περιγράφουμε σε λεπτομέρειες το πώς θα γίνει αυτό. Ζητήθηκε επίσης προσοχή από τους συναδέλφους για το νερό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό φύγει όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία προανέφερα. Στην Ευρώπη, σε, ορισμένα τμήματα της Ευρώπης που υπάρχει πολύ νερό, γίνεται σπα, σπα, σπα, ενώ άλλες χώρες ε, έχουν στην Ευρώπη υπάρχει ξηρασία πρέπει και τεχνολογικά να λύσουμε το πρόβλημα ούτως ώστε να γίνεται μεταφορά. Είναι πάρα πολλές φορές επίσης δύσκολο να έχει κανείς μία σφαιρική εικόνα όλων των διαφόρων προγραμμάτων που, βρίσκουν, που τρέχουν, όλων των αποτελεσμάτων ε, της ε, καινοτομίας. Υπάρχει και κατακαιρματισμός της ίδιας της πολιτικής την οποία αντιμετωπίζουμε σε μια τέτοια φάση κρίσης, αλλά δεν μπορούμε εμείς να επιτρέψουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια του κατακαιρματισμού των κονδυλίων. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τους στόχους μας για την καινοτομία και για την αριστεία. Και σε αυτό εγώ δεν πρόκειται να συμβιβαστώ. Η Κούρβιτς. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή που εργάζεται για εν, εργάστηκε μέσα σε, για ένα ντοσιέ τόσο μακρόπνο. Ο ορίζοντας 2020 είναι ελπίδα για τους πολλούς, είναι ελπίδα και όχι μόνο για τη ιατρική για την υγεία, αλλά και για τους τομείς εκείνους όπου η τα φορά της έρευνας στην καθημερινή ζωή θα οδηγήσει στη δημιουργία μεγαλύτερης απασχόλησης. Εγώ στις τροπολογίες μου που υποστήριξαν και διάφοροι συνάδελφοι αντιμετωπίζω την προπτική της υγείας. Είναι μια προπτική που πρέπει να την έχουμε κατά νου, αλλά λάβει κανείς υπόψη τη γύρανση του πληθυσμού. Να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές τεχνολογίες, μεταξύ των οποίων τις τεχνολογίες μάλλον με τις οποίες ε, επιτρέπεται να σταματήσουν οι ουρές και οι αναμονές ε, στα, για την υγεία. Σίγουρα χρειάζεται ένα υγιεινός τρόπο ζωής, υγιεινή τροφή. Πρέπει να τονιστεί και αυτό να κάνουμε, να κάνουμε σαφές στον κόσμο το τι είναι υγιές διότι η υγεία μας εξαρτάται από το τι απορροφάει ο οργανισμός μας. η νέα γνώση, οι νέες εφευρέσεις, οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής πρέπει να υποστηριχθούν είναι σημαντική και η ταχύτητα αυτών των νέων εφευρέσεων ή νέων προϊόντων, αλλά, πρέπει να, χρειάζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζητώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου. Είμαι πεπισμένη ότι αυτές οι τροπολογίες είναι καλύτερες από όλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόκοβιτς. Γι' αυτό το κάνουμε, για να μπορούν να ωφεληθούν όλοι. Και αυτό υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, να παρακαλέσω την Επιτροπή να σχολιάσει για τα θέματα που τέθησαν. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ τον εισηγητή και τους Σκιώδης και άλλα μέλη της Επιτροπής που έκαναν σημαντική εργασία εδώ. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε ότι η πρόταση της Κομισιό ε, προβλέπει μια συστημική προσέγγιση ε, ε, σχετικά με τους, τα βασικές προκλήσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την προσέγγιση αυτή όσο είναι δυνατόν. Για να διατηρήσουμε αυτή την προσέγγιση και την ευελιξία με το 7 πρόγραμμα ένα μιας μακρύς κατάλογος ιδιαίτερων θεμάτων και λεπτομεριών θα πρέπει να αποφευθεί σε αυτό το στάδιο. Ε, μια, ένας κατάλογος πολύ περιγραφικός μπορεί να έχει ε, μη αναμενόμενες επιπτώσεις σχετικά με δραστηριότητες που θα θέλαμε να εισαγάγουμε σε περαιτέρω στάδιο ως προς τα ειδικά σχόλια για ορισμένα θέματα. Όσον αφορά στην υγεία, στα θέματα υγείας, Βεβαίω, συγχαίρουμε τον εισηγητή για την ευελιξία σχετικά με τα βλαστοκύτταρα και επίσης συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε εδώ πολύ περιγραφικοί όσον αφορά τις εναλλακτικέ επιλογές και το ίδιο ισχύει για το μακρύ κατάλογο αυτών των τεχνολογιών και των ομάδων. Θα θέλαμε επίσης να συμφωνήσουμε με τον ε, εισηγητή όσον αφορά στο θέμα ενός χωριστού κεφαλαίου ε, για την ε, οικολογική καινοτομία. Αυτό δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο, εφόσον το θέμα αυτό καλύπτεται στο 5 στο τμήμα 5, όπου καλύπτεται όχι μόνο όσον αφορά στις τεχνολογίες, αλλά επίσης και όσον αφορά ε, στις ε, κοινωνικές καινοτομίες. Ε, θα πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι το όλο θέμα του ετσαϊφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των θεμάτων του προγράμματος Horizon 2020. Θα πρέπει σε όλα τα τμήματα του προγράμματος αυτού να περιλαμβάνεται, λαμβάνεται υπόψη η αηφόρος ανάπτυξη ως προς το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που τονίστηκε από πολλά μέλη εδώ του ύδατος είναι όντως ε, ήδη ε, καλύπτεται σε διάφορα τμήματα της πρότασής μας. Το να έχουμε ένα χωριστό τμήμα όπως προτάθηκε ίσως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα, διότι το θέμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται σε διάφορα άλλα θέματα, να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, με την διαχείριση υδάτων, με την επεξεργασία υδάτων και υπάρχει και ένα τμήμα που συνδυάζεται με την οικολογική καινοτομία. Σε συνδυασμό με το είδωρο βεβαίως. Υπήρξε επίσης αίτημα για διαφάνεια και συμφωνούμε με αυτήν την πτυχή της διαφάνειας. Γι' αυτό ήδη, ήδη στο 7 υπήρξε ε, το, ένα, μια δυνατότητα ε, ανοιχτής επισκόπησης από μότιμος και αυτό και ήταν μέρος αυτού όλου του σχεδίου και αυτή η όλη προσέγγιση θα προωθηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 και των δραστηριοτήτων του. Τώρα θα ήθελα να πω ως τελευταία παρατήρηση, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, να αναφερθώ στον προϋπολογισμό. Η πρόταση της Κομισιό είναι απόρρια ε, ενό συμβιβασμού ισορροπημένου ανάμεσα στους τομείς πολιτικής που καλύπτει. Ενημερωθήκαμε ότι το NFF του Κοινοβουλίου είναι κατά της συζήτησης του προϋπολογισμού για κάθε τομεακή πρόταση, αλλά εναπόκειται σε εσά να αποφασίσετε. Αλλά βεβαίως σας ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία και θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχείς να συμβάλλουμε στα θέματα τεχνικής βοήθειας για τα διάφορα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Κύριο Μπουζόη, για να αναφερθεί στα ερωτήματα που ετέθησαν από τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κλείστε παρακαλώ το μικροφωνό σας, κύριε της Κομισιόν. Κυρίες της Κομισιόν. Ευχαριστώ, ωραία. Πολύ σύντομο θα είμαι. Πολλοί είπαν πως είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Και πολύ περίπλοκο. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τη συνεργασία της. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία της Επιτροπής μας και τους ε, εμπειρογνώμονες που με βοήθησαν τους προσωπικούς μου εμπειρογνώμονες, τους εμπειρογνώμονες της ομάδας μου που με βοήθησαν λοιπόν. Στην κυρία Κουτιέρεθ Κορτίνεθ. Σημειώνω αυτά που μας είπατε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Όχι, δεν θα αλλάξω τη δομή του προγράμματος. Έχετε υποβάλει πολλές τροπολογίες. Με χαρά θα τις υποστηρίξω. Συμφωνώ βεβαίως ότι είναι σημαντικό το θέμα των υδάτων και βεβαίως όσοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη πρόσβαση. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι για την εξατομικευμένη ιατρική. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι μόνο πολύ φιλόδοξο αλλά εάν επιτύχουμε θα έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικές και οικονομικές θεραπείες άρα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτής της ε, εξατομικευμένης ιατρικής την κυρία Evans την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια Περίμενα ότι οι συνάδελφοί της και εκείνοι θα ασχοληθούν πολύ με την κλιματική αλλαγή. Και για μένα κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα έχουν μεγάλη σημασία. Με αυτό το εργαλείο, καθώς και με άλλα, και με την νομοθεσία θα επιδιώξουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προς την κυρία Ζόουζα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνονται ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι δύο τροπολογίες σας για τα βλαστοκύτταρα περιέχουν ιδέες που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε να βρούμε όλοι μαζί κάποια συμβαστική λύση για αυτό το λεπτό θέμα των βλαστοκυτάρων. Είναι κάτι που ανέφερε και ο συνάδελφος Λίζε. Βεβαίως για την υγεία των ε, παιδιών θα υποστηρίξω τις τροπολογίες του και συνυπέγραψα τις τροπολογίες του για την αντισύλληψη. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της κυρίας Μέρκης ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα σημαντικά θέματα και να μην είμαστε υπερβολικά συγκεκριμένοι, να μην αναφέρουμε πολλές λεπτομέρειες, να μην προτείνουμε πολλά μέτρα. Αυτό το κείμενο θα πάει στην Ήτρα. Να στοχεύσουμε λοιπόν τα σημαντικά θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ και τους συναδέλφους να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε από κοινού σε συμβασμούς όπου είναι εφικτή. Σημερίζομαι το ενδιαφέρον της κυρίας Κόκοβιτς για τον τομέα της υγείας και εγώ είπα πολλά για την υγεία πολλές ιδέες των συναδέλφων είναι ιδιαίτερα πολύτιμες θα αυξήσουν την αξία του κειμένου που προτείνω. Όπως είπα, κατά τις διακοπές μαζί με τους συνεργάτες μου θα προσπαθήσω να καταλήξω σε κάποιους συμβασμούς και προσβλέπω στην συνεργασία μας το Σεπτέμβριο για την επίτευξη σωστών λύσεων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε Μπουζόη, ο Πέτε Λίζε είπε ότι θα πρέπει κάπως να περιορίσουμε τις τροπολογίες, το έλαβα υπόψη. Το είχαμε συζητήσει και προηγουμένως. Θα προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Τώρα βέβαια μέχρι που θα πάμε πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα και που, πώς θα ξεκινήσουμε, πού θα σταματήσουμε. Θα σας ε, ενημερώσω για το τι διαδικασία θα προτείνω. 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια θα περάσει τον Νοέμβριο. Τέλος, να κάνω άλλη μια ανακοίνωση. Ορίστε οι τροπολογίες. Όποιος θέλει άλλη φορά να τις ε, πάρει μαζί του ή να συνεργαστεί, πάρτε τις μαζί σας. Γιατί αν πρέπει να τις ξανατυπώσουμε, είναι 40.000 σελίδε όλες τι γλώσσες. Σας παρακαλώ πάρτε τις. Παρακαλέστε τους βοηθούς σας να πάρουν τα έγγραφα. Γιατί έχουμε γράψει στον εσωτερικό μας κανονισμό ότι θέλουμε να περιορίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Οπότε και ω Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Και περνάμε στο 19. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει 6 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφου για τη συνεργασία μας κατά το πρώτο εξάμεινο. Με βοηθήσατε όπως ανέλαβα την Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γραμματεία και ιδιαίτερα τον κύριο Όβερ για την θαυμάσια υποστήριξη της εργασίας της Επιτροπής μας και όλους τους βοηθούς, όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς γιατί χωρίς τους διερμηνείς δεν θα είχαμε καμία δυνατότητα. Ξεκουραστείτε από εμάς. Και τον Σεπτέμβριο παρακαλώ να έρθετε όλοι πίσω, να επιστρέψετε. Γεμίστε τις μπαταρίες σας. Πολλά καταφέραμε να κάνουμε τους τελευταίους μήνες, αλλά μας περιμένει πολλή δουλειά το δεύτερο ε, μισό του 2012. Σας εύχομαι σε όλους ε, ό,τι καλύτερο, καλές διακοπές.